Je Σας προτείνω να αρχίσουμε τις εργασίες μας, συνάδελφοι. Έχουμε καθυστερήσει κάπως. Σας εύχομαι καλή αρχή. Βλέπω ότι όλοι έχετε μαυρίσει. Έχετε μια ζωηρότητα σε σχέση μεγαλύτερη από εκείνη του Ιουνίου. Άρα ελπίζω να περάσατε ευχάριστες διακοπές με αρκετό αθλητισμό έτσι ώστε όλοι να είμαστε σε φόρμα το φθινόπωρο τούτο του 2011 διότι μας περιμένει το έργο της συζήτησης και της ψήφισης του προϋπολογισμού. Θα αρχίσουν και οι για τις δημοσιονομικές προοπτικές δυστυχώς κάτω από δίκες από πλευράς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Είδατε την ημερήσια διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια θεωρούμε ότι εγκρίνεται. Όπως όσον αφορά τη σειρά της εξέτασης των διαφόρων θεμάτων, στις 10.30 μαζί της ο εισηγητής να ασχοληθούμε με την έκθεση Μπάρμπαρα Ματέρα. Να τη δούμε μεταξύ 10.30 και 11. Τα άλλα θέματα παραμένουν ως έχουν. Και η σειρά ως έχει. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών της 12ης και 13ης Ιουλίου, αν δεν υπάρχουν σχόλια μέχρι το τέλος της συνεδρίασης θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται ως προς τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Υπάρχουν στο κόμπου News, γι' αυτό δεν θα επιμείνω. Η Ντέβε, μαζί με τον κύριο Φιλίππο Γκράντι, από την UNRWA ε, ε, στην Παλαιστίνη, θα έχει να πει πολλά. Είμαστε στο διαδίκτυο και θα ασχοληθούμε και με πρωτίστως μάλλον με την εφαρμογή του προϋπολογισμού 2011. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον Γενικό Διευθυντή Προϋπολογισμών της Κομισιόν, τον οποίο δεν βλέπω στην αίθουσα. Α, όχι, είναι εδώ, είναι εδώ, με συγχωρείτε αλλά κάθισε πίσω-πίσω, όπως οι κακοί μαθητές. Μας θυμάμαι την παρουσία του λοιπόν. Αγαπητή Φραντσέσκα Μπαλζάνη και Ζωζέ Μαλουέρ Φερνάντες, θα αρχίσουμε με τον προϋπολογισμό του 2012. Το καλοκαίρι ενέκρινε με ενιαία ανάγνωση το κείμενο το Συμβούλιο και θα ήθελα να μου πείτε την ε, άποψή σας. Καταρχήν η Φραντσέσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στις 27 Ιουλίου το Συμβούλιο ενέκρινε στην ανάγνωσή του το κείμενο με αντίθετη γνώμη έξι κρατών μελών που δεν ενέκριναν την ανάγνωση του Συμβουλίου θεωρώντας ότι ο προπολογισμός της Ένωσης το 2012 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Και αυτό όχι μόνο όσο αφορά τις πληρωμές, αλλά και τις αναλήψεις υποχρεώσεων. Κατά συνέπεια, η ανάγνωση του Συμβουλίου ήταν μία συσταλτική ανάγνωση σε σχέση με εκείνη της Κομισιόν, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το 2011 είχε προτείνει αύξηση στις υποχρεώσεις 4% και στις πληρωμές 4,9% που μειώνει το Συμβούλιο σε 2,9% και 2% αντιστοίχως υποχρεώσεις και πληρωμές. Το στοιχείο όμως το οποίο είναι πιο χρήσιμο για να καταλάβουμε την παρέμβαση του Συμβουλίου, του Συμβουλίου αφορά το γεγονός ότι πέρα από την μείωση 400 γραμμών το Συμβούλιο δεν έχει αυξήσει ούτε, κα, ούτε καν μία. Πρόκειται λοιπόν για μία ε, μείωση Μεγάλη μείωση. Οι πληρωμές μειώνονται κατά 3 δις 600 εκατομμύρια, ιδιαίτερα τη στήλη 1β οι υποχρεώσεις μειώνονται σε τρεις στήλες, τρία κεφάλαια. Πρόκειται για την 1α, την 2 και τα 4. Η μείωση της 1α αφορά την χρηματοδότηση του Ίτερ, διότι το Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση της Κομισιόν για την χρηματοδότηση με 750 εκατομμύρια και μείωσε σε 650 με βάση τα περιθώρια του 2011, δηλαδή τα ποσά που δεν δαπανήθηκαν. Αντίθετα, επέτρεψε 100.000 100, συγγνώμη, εκατομμύρια από την γραμμή της έρευνες σε ορισμένα προγράμματα όπως η διανομή ε, γάλατος ή οπορεκπαιδευτικών, ιδιαίτερα στα σχολεία, έχουν γίνει μειώσεις. Έγινε μεγάλη συζήτηση στην Κομισιόν με την έγκριση μίας παραγράφου ad hoc. Άρα δέχεται αύξητο το Συμβούλιο κατά 400 εκατομμύρια για την πολιτική γειτονίας, αλλά δεν επιτρέπει την χρήση του μέσου ευελιξίας κατά 150 εκατομμύρια και αφαιρεί πόσα από πολλά μέσα, δηλαδή ανθρωπιστική βοήθεια, μέσο ευελιξίας και ούτω καθεξής. Υπάρχει και το κεφάλαιο 5, στήλη 5, που αφορά τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου όπου γίνονται μειώσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με το προσωπικό, οι δαπάνες προσωπικού. Ως προς τα διάφορα ιδρύματα και εδώ γίνονται περικοπές και επειδή πρόκειται για συγκεκριμένες αζόνς, ιδρύματα ή γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώνονται οι πόροι. Επίσης γίνονται περίκοπες στις δαπάνες, στις διοικητικές δαπάνες, που θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των προγραμμάτων. Άρα το σενάριο αυτό ήταν αυτό της Κόρεπερ στις αρχές Ιουλίου. Δεν έχει διαφοροποιηθεί. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια θα είναι η δική μας στρατηγική σε σχέση με την ανάγνωση του Συμβουλίου, σε σχέση με την Κόρεπερ που είναι το σημείο αναφοράς μας. Ως προς τις πληρωμές καταρχήν. Γνωρίζουμε ότι οι πληρωμές δεν αποτελούν την ψυχή του προϋπολογισμού. Είπαμε ότι οι πολιτικές επιλογές βασίζονται στις υποχρεώσεις και όχι στις πληρωμές. Είναι όμως γεγονός ότι οι πληρωμές μας δείχνουν τι θα συμβεί και με τις υποχρεώσεις. Εάν μιλάμε για πληρωμές που είναι φιλόδοξες και στη συνέχεια το Συμβούλιο δεν μας επιτρέπει να κινηθούμε με τις υποχρεώσεις, στην ουσία μας ε, βγάζει μας ε, αφαιρεί κάθε δυνατότητα παρέμβασης. Ενώ λοιπόν θέλουμε να φτάσουμε σε μια στρατηγική, σε μια πολιτική ως προς τον προϋπολογισμό που βασίζεται στις υποχρεώσεις, εμείς θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να σταθούμε στις υποχρεώσεις γιατί θα ψηφιστούν αύριο και δεν μπορούμε να μελήσουμε και τις πληρωμές διότι ως προς τις πληρωμές είχαμε ψηφίσει και με βάση τον τριμερή διάλογο όπου λέγαμε ότι η πρόταση της Κομισιόν αποτελεί ένα ελάχιστο όρο διαπραγμάτευσης για να μπορέσει ο προϋπολογισμός να είναι πραγματικά λειτουργικός. Και διότι στο τέλος του πακέτου βλέπουμε ότι τα προγράμματα εκτελούνται με καλό ρυθμό. Θα πρέπει λοιπόν να μην υπάρχει αυτό το μεγάλο χάσμα μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών. Προβάλλοντας λοιπόν αυτή τη στρατηγική και επειδή θεωρούμε ότι η Μπαρόζο και Λεβαντόφσκι θα έθεταν έναν ελάχιστο όρο λειτουργικότητας του προϋπολογισμού και μείωση του χάσματος μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών, θα πρέπει να υπεραμεινθούμε αυτή τη θέση της Κομισιόν. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχουν ουσιώδεις αυξήσεις και στις πληρωμές, ιδιαίτερα στη στήλη 1β που πλήττεται ιδιαίτερα. Γιατί χρειαζόμαστε διαθέσιμους πόρους, ιδιαίτερα για τις χώρες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες επενδύσεων. Ως προς τις αναλήψεις υποχρεώσεων, σας είπα ότι αφορούν την 1α, 2 και 4. Αυτές τις στήλες, αυτά τα κεφάλαια. Στην 1α θα πρέπει να δούμε πώς η στρατηγική 2020 θα μπορέσει να επικαιροποιηθεί με βάση τις περικοπές που προβάλλονται. Θα πρέπει λοιπόν να αποκαταστήσουμε την πρόταση της Κομισιόν ιδιαίτερα σε σχέση με τις γραμμές που αφορούν τη στρατηγική 2020. Το ίδιο αφορά και το κεφάλαιο 4 που ασχολείται με τα βασικά στοιχεία που αφορούν την επικαιρότητα, τη λεκάνη της Μεσογείου και την Αραβική Άνοιξη. Αυτό που θα ήθελα όμως, πέρα από την ε, υπεράσπιση αυτών των γραμμών, από θεσμικής πλευράς, που επικαιροποίησε και η Κομισιόν, νομίζω ότι πρωτίστως ως κοινοβούλιο θα πρέπει να σταθούμε σε ιδιαίτερες στρατηγικές και προτεραιότητες. Χρειαζόμαστε έναν περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων για να μην είναι κενές περιεχομένου αυτές οι στήλες, ιδιαίτερα οι επίμαχες. Διότι σε μία περίοδο λιτότητας όπου θα πρέπει να ε, δείξουμε ότι είμαστε συνετοί και ως προς τις δαπάνες, νομίζω ότι πέρα από τις περικοπές θα πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε μια αυστηρή επιλογή των προτεραιοτήτων και να σταθούμε σε συγκεκριμένα θέματα και γραμμές. Όπως η στρατηγική 2020 που είναι και η κατευθυντήρια γραμμή μας κάτι το οποίο δεν τονίζεται στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, να προβούμε σε μια αυστηρή επιλογή προτεραιοτήτων με βάση τα θέματα που είναι ύψη της σημασίας. Ο Ζωζέ Μανουέλ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θα μιλήσω για τον προϋπολογισμό των άλλων θεσμικών οργάνων, καθώς και του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο με βάση μία ε, συμφωνία κυρίων δεν έκανε καμία περικοπή στον ε, προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου. Έκανε όμως περικοπές στα άλλα θεσμικά όργανα. Επίσης, καταβλήθηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τα άλλα θεσμικά όργανα και φορείς και αυτή η προσπάθεια δεν ελήφθη υπόψη από το Συμβούλιο. Ως προς τις αζόνς και τους φορείς, παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να, είμαστε, να προβάλλουμε μια πολιτική λιτότητας, τα ιδρύματα και οι φορείς αυτοί κάναν οι ίδιοι μεγάλες περικοπές. Παρόλα αυτά όμως το Συμβούλιο έκανε επιπρόσθετες περικοπές. Κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχτούμε. Γιατί δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για να καταβληθούν οι δαπάνες, παραδείγματο χάρη ε, του προσωπικού, οι πληρωμές μισθών οι, οι πληρωμές των αναγκών του κτηρίου και ούτω καθεξής. Επίσης, η μελλοντική προσχώρηση της Κροατίας δεν έχει ενταχθεί σε αυτό τον προϋπολογισμό. Σε σχέση με το Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Προϋπολογισμών αναφέρθηκε σε κάθε κεφάλαιο και μιλήσαμε ως προς αυτό το θέμα και στην Ολομέλεια με βάση τις ε, προβλέψεις. Έχουμε λοιπόν μεγάλα ανοιχτά μέτωπα και Σε σχέση με την αρχική πρόταση, εμείς κόψαμε 50 εκατομμύρια και περάσαμε σε μία αύξηση 2,3%. Αυτό προβλεπόταν και ως απότοκο της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα πρέπει λοιπόν να αποσταλεί μία διορθωτική ε, πιστολή για 10 εκατομμύρια 600.000 μετά από την θέση σε ισχύ της συνθήκης. Πρόκειται για τα νέα μέλη, 18 νέα μέλη και αυτό έχει βεβαίως και δημοσιονομικές επιπτώσεις που γνωρίζαμε. Είμαι στη διάθεσή σας και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας. Βεβαίως να μην ξαναρχίσουμε τη συζήτηση για τις προβλέψεις, διότι φτάσαμε σε συμφωνία, αλλά θα ήθελα να ακούσω τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν μεγάλη πείρα, καθώς και τη θέση τους σε σχέση με τους άλλους φορείς και όργανα διότι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν διανύουμε μία εύκολη περίοδο, γι' αυτό θα πρέπει, κατανοούμε, ότι πρέπει να γίνουν περικοπές, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και θεωρούν οι πολίτες ότι θα πρέπει να νομοθετήσουμε καλώς και να λάβουμε υπόψη τις πρωταρχικές ανάγκες των πολιτών. Να μπορέσουμε λοιπόν να ανταποκριθούμε στο έργο μας. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε την ποιότητα ζωής πρωτίστως των πολιτών, γιατί αυτός είναι ο πρώτιστος και ο ίστατος στόχος. Σας ευχαριστούμε κύριε εισηγητά. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές και εισηγήτριες που έκαναν τη δουλειά τους τόσο καλά υπό τόσο δύσκολες συνθήκες. Πρέπει να ξέρουμε όλοι πού βρισκόμαστε και ποιες είναι οι επιλογές μας. Γιατί υπάρχουν επιλογές ως προς τη γενική προσέγγιση αντιμετώπισης αυτής της δύσκολης κατάστασης. Μία θα ήταν να δεχτούμε τη στάση του Συμβουλίου και να ζητήσουμε περικοπάς. Δηλαδή να δεχτούμε μια ελάχιστη γραμμή με βάση τα επιχειρήματα που εκφράζουν οι χώρες μέλη κλπ. Αυτή είναι μία επιλογή. Τέπει τουλάχιστον να τη συζητήσουμε. Δεν είμαστε υπέρ, αλλά να τη συζητήσουμε. Άλλη επιλογή θα ήταν η συνήθις, δηλαδή να επαναφέρουμε το προσχέδιο προϋπολογισμού της Κομισιόν και να στηρίξουμε έτσι την Κομισιόν. Τρίτη επιλογή θα ήταν να είμαστε πολύ ριζοσπαστικοί και να πούμε ότι δεν δεχόμαστε τη λιτότητα και θέλουμε ριζική αναθεώρηση των προοπτικών κλπ. Και τέταρτη επιλογή που είναι και αυτή που θα υποστηρίξουμε εμείς είναι μια επιλεκτική προοπτική δηλαδή μερικές ριζικές αυξήσεις αλλά σε πολύ συγκεκριμένους και πολιτικά σημαντικούς τομείς όπως το πρόγραμμα 2020 και ιδιαίτερα τα τμήματά του που αφορούν την ανάπτυξη και την απασχόληση όπως τη διαβίωμάθηση, ε, έρευνα κλπ. Άλλο παράδειγμα στην κατηγορία 4, σε ένα τμήμα της κατηγορίας 4 όπως τα νέα εργαλεία για την καλή γειτονία και τι πρέπει να γίνει για τον νότο της Μεσογείου. Αυτή είναι η γενική μας άποψη. Δεν θέλουμε επαναφορά όλων των κονδυλίων. Δεχόμαστε μερικές από τις ε, περικοπές του Συμβουλίου, όχι όλες μερικές, αλλά σε επίλεκτους τομείς όπου θεωρούμε ότι υπάρχει τεράστια πολιτική προτεραιότητα είμαστε προετοιμασμένοι να δώσουμε σκληρό αγώνα. Αυτή νομίζω είναι η καλύτερη στάση, αλλά πρέπει βέβαια να αναλύσουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Όχι μόνο να καθορίσουμε πολιτικές προτεραιότητες, αλλά να δούμε και ποια δυνατότητα υπάρχει εφαρμογής τέτοιων αυξήσεων που θα ζητήσουμε. Η Φραντσέσκα μας είπε από την αρχή ότι η δική της στάση βασίζεται στο δημοσιονομικό πρόγραμμα που έχει εκφραστεί. Πρέπει όμως να δούμε ποιες από τις ανάγκες που αναφέρει μπορούν να εφαρμοστούν ως αυξήσεις. Αυτή είναι η κυρία δουλειά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Με τις πολιτικές λοιπόν προτεραιότητες, τις δυνατότητες εφαρμογής και απορρόφησης νομίζουμε ότι θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε μια στρατηγική που να είναι εφαρμόσιμη αλλά και εξηγήσιμη προς το ευρύτερο κοινό. Αυτή είναι η βασική μας τάση. Η Φραντσέσκα λέει ότι οι προβλέψεις είναι σημαντικότερες από τις πληρωμές. Ναι, πολιτικά ναι, αλλά πρέπει να γίνει μια πραγματική συζήτηση και για τις πληρωμές διότι οι πληρωμές θα δημιουργήσουν την ανάπτυξη επιτόπου που είναι αυτό που θέλουμε αυτή τη στιγμή. Οι προβλέψεις είναι απλώς πολιτικές υποσχέσεις ενώ η πραγματικότητα είναι οι πληρωμές. Πρέπει να συζητήσουμε και μερικές πληρωμές λοιπόν. Για τα άλλα όργανα Κατανοούμε τι θέλει το Συμβούλιο. Δεν είναι ποτέ εύκολο να διατηρηθεί μια καλή διοίκηση υπό δύσκολες συνθήκες, αλλά νομίζω έχουν ξεπεράσει τα όρια. Δηλαδή εμποδίζουν την εργασία βασικών οργάνων. Όχι απλώς εξοικονομήσεις ζητούν, αλλά ζημιώνουν τη λειτουργία τους. Και αυτό δεν είναι σωστό. Και εδώ νομίζω πρέπει να είμαστε επιλεκτικοί. Να δεχτούμε μερικές από τις εξοικονομήσεις, δηλαδή περικοπές, αλλά να προσπαθήσουμε να διατηρηθεί η βασική δουλειά των οργάνων. Αλλιώς θα δημιουργηθούν νέα προβλήματα στην εφαρμογή. Και Τέλος, για τον δικό μας προϋπολογισμό του κοινοβουλίου δηλαδή. Ο δικός μας είναι ο μόνος προϋπολογισμός που δεν είναι ο μόνος που έχει περικοπεί από το Συμβούλιο. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε το δικό μας θα τον επαναφέρουμε αλλά τους άλλους, των άλλων οργάνων άσκοπου είναι οι προϋπολογισμοί. Πρέπει να βρούμε και εμείς πρόσθετες εξοικονομήσεις υπάρχει τρόπος χωρίς να βλαφτεί η λειτουργία του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι πολιτικά κάτι τέτοιο είναι απολύτως απαραίτητο. Ευχαριστούμε Γκέραν ο κύριος Λαβίας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι καταρχήν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τους δύο συντάχτες, Μπαλζάνη και Φερνάντες, για την ε, εξαιρετική παρουσίασή τους και γιατί μας ε, επέστησαν την προσοχή σε συγκεκριμένα θέματα. Υπάρχει ένα πρώτο θέμα που αφορά τις επιλογές μας για να δούμε σε μια περίοδο κρίσης κατά πόσο είμαστε αρκετά φιλόδοξοι. Δηλαδή, διανύοντας αυτή τη δύσκολη περίοδο, κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ε, πραγματικές και ρεαλιστικές ανάγκες κατανοώ ότι σε μία περίοδο κρίσης που διανύουμε, που φάνηκε με τις έξι, από τις έξι χώρες που αντιτάχθηκαν στην υπέρβαση του ε, πληθωρισμού, δηλαδή ε, στην υπέρβαση του τιμαρίθμου, δείχνει ότι πραγματικά διανύουμε μια μεγάλη κρίση που αντικατοπτρίζεται σε πολλές χώρες. Αλλά μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών, γιατί διανύουμε το πρώτο τελευταίο έτος, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες. Δηλαδή να είμαστε επιλεκτικοί. Και ο προϋπολογισμός θα πρέπει να μπορέσει να ορίσει τις γραμμές που αποτελούν προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο, γιατί οι περικοπές δεν είναι κατανοητές, τουλάχιστον όλες οι περικοπές του Συμβουλίου. Γιατί η στρατηγική 2020 διαβίου μάθηση, η ΜΜΕ στο κεφάλαιο 1α περικόπτονται, ενώ θα έπρεπε να τύχουν υποστήριξης για να μπορέσουμε σε μία περίοδο κρίσης να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Επίσης, το 3α γίνονται περικοπές ως προς τα προγράμματα της ε, Μεσογείου, τη Frontex, το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Πρόκειται για περικοπές οι οποίες είναι άνευ νοήματος και νομίζω ότι θα πρέπει να αντιταχθούμε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αξιολόγηση που να λαμβάνει υπόψη προτεραιότητες οι οποίες ορίζονται σαφώς και να ζητήσουμε την ανάκτηση των αρχικών μας προτάσεων και ποσών όπως είχαν προταχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι διανύουμε αυτή τη μεγάλη περίοδο κρίσης και θα πρέπει να ε, δώσουμε εμείς την προστιθέμενη αξία των προτάσεων. Και γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε στοχοθετημένες προτάσεις με σαφή μηνύματα. Αυτά, αυτό θα πρέπει να είναι το κεντρικό μας μήνυμα προς την Ευρώπη. Αν Γένσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τους συζητητές για τις πολύ σαφές εξηγήσεις που μας έδωσαν. Θα έλεγα ότι η Άλντε πιστεύει ότι ασφαλώς και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εξετάσουμε γενικά πώς έχει η κατάσταση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι δαπάνε δεν θα είναι πιο υψηλέ από τα βασικά απαιτούμενα. Και γι' αυτό σύμφωνο με την γραμμή των σοσιαλιστών και με αυτά που μας είπε ο κύριος Λαβία, ότι θα πρέπει να θέσουμε αυστηρές προτεραιότητες σε ό,τι αφορά την αύξηση του προϋπολογισμού σε σχέση με τα επίπεδο που προτείνει το Συμβούλιο να πω ότι ακόμα και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάποιους τομείς θεωρούμε ότι ήταν αρκετά σφιχτή. Και κάποιες εξωτερικές υπηρεσίες, ε, οργανισμοί θα έχουν προβλήματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι πολύ λεπτομερής η ανάλυση μας. Γιατί βλέπουμε ότι γίνονται και πάλι περικοπές πολύ περίεργες ε, σε σχέση και με τις προτεραιότητες που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για παράδειγμα, γιατί γίνονται περικοπές στην Αραβική Άνοιξη, στον Frontex, όλα αυτά μας φαίνονται πολύ περίεργα. Επίσης γνωρίζω ότι υπάρχουν και διαφορές στο εσωτερικό του Συμβουλίου και ξέρω ότι κάποιες χώρες καταψήφισαν τις προτάσεις του Συμβουλίου γιατί θεωρούν ότι για παράδειγμα οι περικοπές στην έρευνα είναι υπερβολικές και είναι υπερβολικέ. Συμφωνώ. Αυτό είναι αντίθετο με τη στρατηγική το 2020 και δεν θα πρέπει να το αποτεχτούμε σε καμία περίπτωση. Να κοιτάξουμε τομεί όπου θέλουμε να μην γίνουν περικοπές ή που θέλουμε ίστως να γίνουν και αύξηση του προπολογισμού. Έγινε και συζήτηση για τις πληρωμές και τις υποχρεώσεις. Νομίζω ότι βλέπουμε πλέον ότι οι υποχρεώσεις είναι για το Κοινοβούλιο και οι πληρωμές είναι για το Συμβούλιο. Βλέπουμε να επιβεβαιώνεται αυτό το παλιό ρητό. Αλλά τι βλέπουμε επίσης σήμερα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταφέρει χρήματα στις αρχές του έτους από προγράμματα που δεν ξέρουμε κατά πόσον θα μπορούσαν να συνεχίσουν. Μεταφέρονται λοιπόν κονδύλια σε άλλα προγράμματα. Άρα έχει σημασία το κατά πόσον έχουμε τα σωστά αριθμητικά στοιχεία για τις πληρωμές, γιατί ιδάλλως δημιουργούμε επιπλέον προβλήματα και αν περιμένουμε ότι το Συμβούλιο θα δώσει επιπλέον χρήματα, να το ξεχάσουμε γιατί δεν πρόκειται να συμβεί. Και θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε και τις πληρωμές και την πλευρά των πληρωμών. Και συμφωνώ ότι οι προτεραιότητες θα είναι στο 1α στην πολιτική εξωτερικών υποθέσεων και θα πρέπει να γίνει ε, να μην γίνει περικοπές. Κάτι περίεργο γίνεται τώρα στη γεωργία, στην εκαθάριση των λογαριασμών για να γίνουν ε, αποταμιεύσεις. Να το κάνουμε μεν, αλλά όχι με τόσο άστοχο τρόπο, λίγο πιο έξυπνα κάποιοι από την ομάδα μου θα προσπαθήσουν να γίνουν περιττέρω περικοπές στα δραστατικά ταμεία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συμφωνήσει η ομάδα μας καν, πόσο μάλλον αν θα συμφωνήσει και όλο το, το Κοινοβούλιο. Αλλά το επιχείρημά μας είναι το εξής. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις, έχουμε ένα τεράστιο όγκο κονδυλίων για τα διευθυντικά ταμεία. Κάποιε από αυτές τις δεσμεύσει θα θέλαμε να τοποθετηθούν στο αποθεματικό και να λάβουμε κάποια εξήγηση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για το τι θα κάνουν με, το, με τα κονδύλια αυτά. Έχουμε 200 ε, δισεκατομμύρια ευρώ σε δεσμεύσει. Τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα αυτά. Θα αποδεσμευθούν κάποια από τα χρήματα αυτά. Τι θα γίνει, εν πάση Κατά δεύτερον, για τις πληρωμές. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου κάποια κράτη-μέλη δυσκολεύονται να εκτελέσουν τα έργα, τα project των διαστατικών ταμείων τους λόγω εγχώριων προβλημάτων των εθνικών δημοσιονομικών τους. Και το... Είναι μόνο μια εκτίμηση σε ό,τι αφορά τις... Γίνεται μόνο μια εκτίμηση σε ό,τι αφορά τις πληρωμές. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι είναι υπερβολικά υψηλή αυτή η εκτίμηση. Αν θέλουμε να περιορίσουμε τις πληρωμές, ίσως καλύτερα να τις περιορίσουμε εδώ. Να μην τις περιορίσουμε τις πληρωμές στο 1α και όχι να μην τις περιορίσουμε και στο 4 και να προσέξουμε, θεωρώ, και την κατηγορία 3. Merci, Anne. Elga η Γέλικα Τρίπελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με τα τέσσερα σενάρια που ανέφερε ο Γκέραν. Είπε ότι όλα θα πρέπει να τα συζητήσουμε, ακόμη αν και αυτός προτιμάται το τέταρτο. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε όλα. Θεωρώ ότι πιο πολύ θα άξιζε να κοιτάξουμε την πραγματική μας στρατηγική. Γιατί αν αποδεχτούμε την θέση του Συμβουλίου θα ήταν πάρα πολύ περίεργα όλα όσα κάναμε ως τώρα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όλα όσα ψηφίσαμε θα ήταν πολύ περίεργα. Άρα δεν πιστεύω ότι είναι ρεαλιστική ε, αυτή, αυτό το σενάριο και δεν θέλω να το συζητήσουμε. Για το τέταρτο σενάριο θεωρώ ότι είναι ο καλύτερο τρόπο αντιμετώπιση τη κατάσταση. Γιατί αυτό που μα παρουσίασε το Συμβούλιο θεωρώ αυτή η αύξηση είναι στα επίπεδα του πληθωρισμού. Είναι πολύ αυστηρή. Αυτό που θέλουν είναι καλύτερη διαχείριση, σύμφωνη ως έναν βαθμό, γιατί η καλή οικονομία προαπαιτεί μια καλή διαχείριση και φυσικά ζητούν και ε, περικοπές και χρησιμοποιούν ένα πολύ δημοφιλές επιχείρημα ότι πρέπει να κάνουμε περικοπές στα κράτη-μέλη Άρα το ίδιο απαιτείται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το γενικό επιχείρημα και σε αυτό το επιχείρημα θα πρέπει να ανταποκριθούμε. Αυτό είναι το βασικό μας καθήκον, θεωρώ. Έγινε μια συνάντηση με τους Γερμανούς πρεσβευτές στο Βερολίνο και καλέσαμε και ένα Γάλλο, έναν Ούγγρο και ένα Πολωνό. Α, και είναι Βρετανό. Και ήταν σαφές το ότι εκτιλήσεται σήμερα στο Συμβούλιο. Είναι μια ιστορία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε. Και λένε ότι θέλουν καλύτερη διαχείριση, αλλά εκ παραλίλου λένε ότι ναι, εγώ θέλω όμως την Βρετανική έκπτωση να διατηρηθεί. Και φυσικά πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολλά, αλλά σε εθνικό επίπεδο δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα και μόνο τα εθνικά, εγωιστικά του συμφέροντα τους απασχολούν. Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα με το οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι. Άρα το ερώτημα που ανακύπτει είναι τι θα κάνουμε. Καταρχάς αυτό που είπε η Αν υπάρχουν και εσωτερικέ διαμάχες, θα πρέπει να τις αξιοποιήσουμε, γιατί μεταξύ των καθαρών ε, ε, εισφορέων και των άλλων χωρών υπάρχουν φυσικά αντικρουόμενα συμφέροντα. Το θέμα είναι Ποια συμφέροντα επικρατούν. Τι θέλουν οι χώρες που λαμβάνουν, για παράδειγμα, κονδύλια και κατά πόσον αυτό αποτελεί την προτεραιότητά μα. Δεν ξέρω. Ύστερα. Τι άλλο έχουμε να κάνουμε. Να καταστήσουμε σαφέ σε πολιτικό επίπεδο ποιο είναι το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον για να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, να κερδίσουμε σε επενδύσεις, σε θέσεις εργασίας, να ακολουθήσουμε τους, τους στόχους της στρατηγικής του 2020. Γιατί αυτό θα πρέπει να είναι το κοινό συμφέρον μεταξύ Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Αυτά έχουμε συμφωνήσει από κοινού. Το ερώτημα είναι, προτίθενται να ακολουθήσουν αυτές τις πολιτικές νέων επενδύσεων. Και γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω την γραμμή του Γκέρεν τις καλές και βιώσιμες δημόσιες επενδύσεις σε ευρύ φάσμα, σε στην έρευνα και την ανάπτυξη, στην ε, εκπαίδευση, όλα όσα καλύπτονται από την ταμπέλα, αν θέλετε, της καινούργιας ανταγωνιστικότητας για την Ευρώπη του 2020 και αφετέρου, όντως αληθεύει ότι σε ό,τι αφορά την κατηγορία 4 και με την Αραβική Άνοιξη, είναι κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον αυτά που διακήρυξε το Συμβούλιο και πάλι. Άρα θεωρώ ότι υπό τις παρούσες πολιτικές συνθήκες η μοναδική ευκαιρία που έχουμε είναι να τονίσουμε τα κοινά ευρωπαϊκά συμφέροντα, το πώς θα πρέπει να ανταποκριθούμε στα κοινά ευρωπαϊκά προβλήματα και ναι, ότι ω ένα βαθμό πρέπει να ακολουθήσουμε την οδό τη λιτότητα, αλλά δεν είναι αυτή η μοναδική απάντηση, όπω βλέπουμε και στην Ελλάδα και σε άλλε χώρε. Χρειαζόμαστε ένα συνδυασμό λιτότητα σε κάποιου τομεί και επενδύσεων, καθαρών επενδύσεων σε άλλου τομεί. Και ελπίζω αυτό να το κατανοήσουν και οι πολίτε, γιατί και τα δικά του συμφέροντα προκύπτουν από τη νέα αυτή ανταγωνιστικότητα. Αυτή θα ήταν η δική μου γραμμή για την επιχειρηματολογία μα. Merci Elga, c'était très clair. James Uh, uh, um, Ευχαριστώ πολύ, Άλαν. Εγώ δεν μπόρεσα να διαβουλευθώ με τους συναδέλφους της ομάδας μου και γι' αυτό θα πω την προσωπική μου άποψη στη σημερινή συζήτηση. Μέχρι σήμερα η ομάδα μου γενικά ακολουθούσε τη γραμμή του παγώματος των αυξήσεων όπως γινόταν και όπως κάναμε και πέρυσι. Αλλά τώρα θα ήθελα να συμφωνήσω λίγο περισσότερο από, με τους προηγούμενους ομιλητές, ιδιαίτερα με τον Γκόραν Φέρμ, διότι νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια διεθνή συγκυρία όπου δεν υπάρχουν πολλοί πόροι, τεράστια χρέη και η προοπτική να μας χρηματοδοτήσει τα χρέη Κίνα δεν είναι πολύ ελκυστική. Πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε προτεραιότητες για να δούμε πού θέλουμε να βάλουμε χρήματα και πού όχι. Αυτή είναι η μόνο, μόνη λογική στάση γιατί αφού υπάρχει και η στρατηγική του 2020 ξέρουμε τι έχει συμφωνηθεί ως προτεραιότητες και σε αυτά πρέπει να επικεντρωθούμε και αφού στις δυτικές τουλάχιστον χώρες συζητιέται το θέμα του κατά πόσον πρέπει να ληφθούν υπόψη μέτρα ενίσχυση της απασχόλησης πρέπει να δούμε να δώσουμε έμφαση κυρίως στην ανάπτυξη πρέπει να βρούμε λοιπόν κάποια κίνητρα και κάποια όθηση για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του κόσμου στο οικονομικό του μέλλον. Επίσης, όπως είπε και ο Γκόραν, πρέπει κυρίως να επιλέξουμε τι ακριβώς είναι εφαρμοσιμότερο γιατί δεν θα άξιζε τον κόπο να κάνουμε προτάσεις και τελικά και εκ των υστέρων να ανακαλύψουμε ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν. <clears throat> Δεύτερο στοιχείο που δεν το έχουμε σκεφτεί αλλά το είπε Φραντσέσκα είναι ότι μπορούν να γίνουν εξοικονομήσεις υπάρχουσες θέσεις αλλά πρέπει πρώτα να γίνει ολόκληρη ανάλυση. πού μπορούν να γίνουν εξοικονομήσεις στα υπάρχοντα προγράμματα. Το καλοκαίρι προσπάθησα να θέσω 60 ερωτήματα στην Κομισιόν <clears throat> για να δούμε πού έχουν χορηγηθεί υψηλά ποσά πάνω από 10 εκατομμύρια χωρίς να έχουν απορροφηθεί. Καταλήγουμε έτσι σε εξοικονομήσεις πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι καλύτερη μέθοδος από τις τυχαίες σχεδόν περικοπές που κάνει το Συμβούλιο που καταλήγουν τελικά στο να μην μπορούν να εφαρμοστούν ορισμένες συγκεκριμένες θέσεις του προϋπολογισμού. Η εξοικονόμηση λοιπόν χρημάτων πρέπει να γίνεται χωρίς να επηρεάζονται και να βλάπτονται οι κύριες θέσεις και προγράμματα που έχουμε εγκρίνει. Τέλος για το προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου και εκεί κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει. Είπε ο Γκόρα να δούμε πού μπορούν να γίνουν εξοικονομήσεις στον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Δεν νομίζω ότι θα προταθούν ποτέ περικοπές στις απολαβές των βουλευτών αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνουν περικοπές ούτε για θέματα πολυγλωσσίας αλλά θα μπορούσαν να γίνουν περικοπές γενικότερα στη διοργάνωση όπου αυτή τη στιγμή ζητούμε να έρχονται διερμηνείς από πολύ μακριά για να εξυπηρετήσουν καμιά φορά γλώσσες που δεν μιλούν σε συνεδρίαση. Ο τωρινός προϋπολογισμός του Κοινοβουλίου στον τωρινό προϋπολογισμό περίπου 50% δαπανάται για τις μεταφράσεις και τη διερμηνία. Χωρίς λοιπόν να βλάψουμε την αρχή του, της πολυγλωσσίας θα μπορούσαμε εκεί να κάνουμε οικονομήσεις εκατομμυρίων. Ευχαριστούμε James. Πάλι Βρετανός αλλά σοσιαλιστός, ο Ντέρεκ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα τους προβολισμούς των άλλων οργάνων. Πρώτα όμως να σχολιάσω την πρόταση των φιλελευθέρων ότι μπορούν να γίνουν περικοπές στα διαρθρωτικά μας ταμεία. Αυτό νομίζω ότι δεν θα ήταν σοφό πολιτικά, ούτε οικονομικά, γιατί πρέπει να προσπαθήσουμε να βάλουμε χρήματα στην απασχόληση και την ανάπτυξη, άρα στα διαρθρωτικά ταμεία. Είναι λοιπόν και πολιτικά μη σοφό να γίνουν εκεί περικοπές γιατί στο μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας της Ένωσης εκεί είναι οι πιο ορατές δαπάνες για τον κόσμο. Να περικοπούν λοιπόν αυτές θα ήταν και πολιτικά λάθος. Τώρα για τα άλλα όργανα. Ευχαριστώ τον εισηγητή κ. Φερνάντες για όσα έκανε για αυτό το θέμα, αλλά και για τη στάση του γενικότερα. Το Συμβούλιο λοιπόν προτείνει περικοπή στους διοικητικούς προλογισμούς σχεδόν όλων των οργάνων εκτός από το Κοινοβούλιο λόγω της περίφημης συμφωνίας κυρίων. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έχει αύξηση κατά 2,3% του προϋπολογισμού του που την είχαμε εγκρίνει στο Προεδρείο μετά από δύσκολες συζητήσεις, αλλά το θέμα τώρα που τίθεται είναι δεχόμαστε και τώρα αύξηση 2,3% ή όχι. Μπορεί οι συνάδελφοι να θέλουν να δουν μήπως πρέπει να γίνουν αυξήσεις σε προϋπολογισμούς και άλλων οργάνων. Το Συμβούλιο παραδείγματο χάρη περικόπτει κατά 5,4% τον προπολογισμό του και η Κομισιόν αυξάνει τον δικό της μόνο κατά 0,4%. Πρέπει λοιπόν και εμείς να σκεφτούμε μήπως πολιτικά δεν θα ήταν φρονιμότερο να κάνουμε και εμείς μερικές επιλεκτικές περικοπές ε, εξοικονομής ενεργείας λοιπά Ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολο μετά από τις συζητήσεις που κάναμε στο Προεδρείο αλλά πρέπει να κάνουμε κάποια προσπάθεια να ταυτίσουμε ορισμένες επιλεκτικές εξοικονομήσεις εμείς οι σοσιαλιστέ θα καταθέσουμε σχετικές προτάσεις. Για τα άλλα όργανα λοιπόν πάλι, όπως είπε ο κύριος Φερνάντες, το Συμβούλιο προτείνει περικοπές ιδίω ως προς τα ναύλα τους και τις, τα έξοδα για τις μεταφράσεις. Σε μερικά όργανα 2,9% και για το ΕΚΟΣΟΚ όχι αύξηση 1,5% αλλά περικοπή 0,5% πράγμα το οποίο θα καταστήσει πολύ δύσκολη τη λειτουργία του. Πρέπει λοιπόν να επαναφέρουμε μερικές θέσεις από τους προλογισμούς των άλλων οργάνων, όχι όλες, αλλά να μπορούν να λειτουργούν όπως πρέπει. Και πάλι θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Μια μικρή αυξησούλα στους προπολογισμούς των Ευχαριστούμε, Σαλβαδόρ Γαρίγα. Πρόεδρε, μερικά από τα σχόλια συναδέλφων θα πρέπει να αποτελέσουν ε, βάση αποφάσεων. Βρισκόμαστε στο δεύτερο έτος εφαρμογής της συνθήκης της ε, Λισαβόνας σε δημοσιονομικά θέματα και βλέπουμε ότι πρέπει να πάμε στη διαδικασία συνδιαλλαγής άμεσα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρά προσκόμματα. Δεν θα πρέπει να έχουμε μονομερή δήλωση από πλευρά Συμβουλίου ως προς το επίπεδο των πληρωμών όπως έγινε πέρσι. Επίσης, το 2012 θα είναι το χειρότερο έτος για τα κράτη-μέλη ως προς τα δημοσιονομικά τους και αυτό αφορά τις περικοπές στους εθνικούς προϋπολογισμούς, κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και στον κοινοτικό. Βεβαίως είναι περίεργη η ανάγνωση του Συμβουλίου που ε, θέτει τις πληρωμές σε διαφορετικό επίπεδο από τις αναλήψεις υποχρεώσεων, το οποίο σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρει να υπάρξει αντιστήχηση. Επίσης δεν υπάρχει αυτόνομο σύστημα ίδιων πόρων, αυτοκυρίαρχο σύστημα ίδιων πόρων, το οποίο σημαίνει ότι τελικά θα επικρατήσει η θέση του Συμβουλίου μετά τη συνδιαλλαγή. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει νέο χρήμα μέσα στα πλαίσια και του μέσου ευελιξίας. Για πρώτη φορά φέτος η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να προβεί σε μία ιεράρχηση σε μια σαφέστερη ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Γι' αυτό οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να συμφωνήσουν ως προς τις προτεραιότητες αυτές, να δουν δηλαδή τι θα δεχτούν ως προς τα προγράμματα, τα οποία έχουν αυξηθεί. Να δούμε ποια προγράμματα και μέσα είναι σημαντικά για μας. Αυτό αφορά και τα flagships της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020. Και νομίζω ότι στο τέλος θα πρέπει να προβούμε σε μια πιο πολιτική ανάγνωση σε σχέση με προγενέστερα χρόνια. Επίσης, φέτος δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου ως προς τον δικό μας προϋπολογισμό βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Δεν είναι λογικό άλλα ε, θεσμικά όργανα και οργανισμοί να κάνουν περικοπές πάνω από τον προϋπολογισμό και εμείς να ακολουθούμε ανωδική πορεία. Θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό μας σε ε, ένα συν 2%. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα ε, επαρκέσει ως προς τους οργανισμούς και υπηρεσίες μας. Θα πρέπει ίσως να γίνουν περισσότερες περικοπές, διότι αυτό είναι το χειρότερο δημοσιονομικό έτος και ίσως θα πρέπει να προβούμε και σε περαιτέρω περικοπές. Θα πρέπει λοιπόν και με τους εισηγητές μας να δούμε πού μπορούμε να κάνουμε περικοπές έτσι ώστε να έχουμε ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί αλλού. Τα αμπάντα. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ce qui a été dit jusqu'à maintenant, je crois que euh, on voit bien qu'on est dans une période extrêmement. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο ο προϋπολογισμός μας μας επιτρέπει να προσδώσουμε προστιθέμενη αξία σε ορισμένα προγράμματα. Γι' αυτό θα πρέπει να στοχοθετήσουμε τις προτεραιότητες. Και εγώ λυπούμε για περικοπές που έγιναν εδώ και εκεί, ιδιαίτερα ως προς τη Frontex, καθώς και τα προγράμματα της διαστημικής μας πολιτικής. Μιλήσαμε για υπηρεσίες και οργανισμούς που διανύουν μία περίοδο κρίσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι μειώνονται οι πιστώσεις τους. Θα πρέπει όλες οι πολιτικές ομάδες να ορίσουμε αυτές τις προτεραιότητες και να δούμε κατά πόσο βελτιώσουμε, μπορούμε να βελτιώσουμε λίγο την κατάσταση. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα πρέπει να δει πού ακριβώς πρέπει να γίνουν οι περιχωπές. Επίσης ένα άλλο θέμα είναι ότι θα πρέπει να πιέσουμε διάφορους οργανισμούς. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Βοήθεια στους πλέον ενδεείς είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν διαθέτει νομική βάση. Θα πρέπει λοιπόν να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη ή στα θεσμικά μας όργανα, έτσι ώστε να μπορέσει να ενταχθεί και να μην πληγεί τόσο πολύ, διότι αυτό προβάλλει αρνητική εικόνα για μας. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μία εξισορροπημένη πρόταση. Εγώ Ήθελα να αποφύγουμε μεγάλες αυξήσεις του προϋπολογισμού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθούμε στο άλλο άκρο. Θα πρέπει να βρούμε, να βρούμε μία εξισορρόπηση, να δούμε ποιες είναι οι βασικές γραμμές δαπανών. Ξέρουμε ότι το κόστος της μετάφρασης είναι πολύ υψηλό. Εάν δεν θέλουμε να πλήξουμε την πολυγλωσία, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά τις υπηρεσίες μεταφο... μετάφρασης και διερμηνίας. Δηλαδή, να μην έχουμε συγκέντρωση συνεδριάσεων μόνο Τρίτη και Τετάρτη, αλλά να υπάρχει μία σωστή κατανομή. Δηλαδή, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, έτσι ώστε να γίνει καλύτερη κατανομή και των υπηρεσιών διερμηνίας. Και επίσης ως προς το καθεστώς των βουλευτών δεν νομίζω ότι θα πρέπει να επέλθουν άλλες ανάγκες, άλλες αλλαγές, με συγχωρείτε. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς μπορούμε να εντάξουμε καλύτερα τις αρχές της συνθήκης της Λισαβόνας στον προπολογισμό. Όπως είπε και ο Σαλβαδόρ, σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Αλλά οφείλουμε να ορίσουμε προτεραιότητες. Διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε ένα σύστημα ίδιων πόρων. Αν δεν έχουμε ένα τέτοιο σύστημα θα είναι πολύ δύσκολο να διαπραγματευόμαστε με τα διάφορα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος Λαμασούρ. Κλείνει η συζήτηση. και βλέπω ότι υπάρχει σύγκληση απόψεων μεταξύ των ομάδων. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που είναι πολύ πιο δύσκολη από την περισσυνή, διότι από πλευράς Συμβουλίου έχουμε δύο κατηγορίες χωρών. Χώρες που γνωρίζουν μεγάλες δημοσιονομικές δυσκολίες και χρειάζονται την στήριξη των εταίρων τους ε, και από τις οποίες δεν μπορούμε να ζητήσουμε αύξηση της συνεισφοράς στον κοινοτικό προϋπολογισμό και απ' την άλλη έχουμε χώρες που πρέπει να χρηματοδοτήσουν τις χώρες που βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι το εθνικό του κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει αυτές τις αποφάσεις. Εδώ μιλώ για τις χώρες της Ευρωζώνης, δηλαδή πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο η βοήθεια προς τις πλέον ενδεείς χώρες και ξέρουμε τι προβλήματα τίθενται. Κατανοούμε ότι η θέση του Συμβουλίου είναι πολύ πιο δυσμενής από την Περσίνη. Από την άλλη πλευρά διαπιστώνω ότι αυτό που είπε ο Γκέραν, η επιλογή υπαριθμών 4, η επιλογή 4 μπορεί να γίνει αποδεκτή από πολλούς δηλαδή μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ορισμένες προτεραιότητες με βάση την Ευρώπη 2020 και τις ανάγκες, την ανάγκη του να ξαναβρούμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής πειθαρχία. Αυτός είναι και ο τετραγωνισμός του κύκλου για τον οποίο μιλάμε εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με το δικό μας προϋπολογισμό. Ζήτησα από τον Αντιπρόεδρο Πιτέλα να προσέλθει να σας παρουσιάσει τις τελευταίες προτάσεις της διάσκεψης προέδρων του Προεδρίου μετά από τη συζήτηση για την Κροατία τη συζήτηση που θα γίνει στο Συμβούλιο. Και τέλος, και μια πιο εύθυμη νότα. Το 2,92% είναι ο μαγικός αριθμός του Συμβουλίου. Πέρσι τον ψήφισαν για τις πληρωμές, φέτος τον ψήφισαν για τις υποχρεώσεις. 2,92%. Βεβαίως θέλει να περιορίσει το Συμβούλιο τις ε, ε, πληρωμές στο επίπεδο του πληθωρισμού. 2,02% προβλέπεται από την Κομισιόν, ίσως να είναι και λίγο ανώτερος ο πληθωρισμός. Λοιπόν, σας προτείνω, οι εισηγητές άκουσαν τι ελέγχθη, δεν θα τους ξαναδώσω το λόγο, αν δεν το επιθυμούν διακαώς. Σας υπενθυμίζω ότι Όσον αφορά τις προθεσμίες μας, έχουμε την, την 8 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σήμερα στις 12 το μεσημέρι, οι επιτροπές που σχετίζονται με το προϋπολογισμό έχουν την ε, προθεσμία αυτή. Οι πολιτικές ομάδες στις 15 Σεπτεμβρίου, την επόμενη εβδομάδα, και η ψηφοφορία Μάλλον θα, ξαναψηφί... θα ξαμιλήσουμε για τον προϋπολογισμό στις 20 Σεπτεμβρίου και στις 4, 5 και 6 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Ωραία, σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο σημείο 4. Όχι, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Ο point 5 l'ordre du 5. όχι, όχι, το είπαμε αυτό, το Περνάμε λοιπόν τώρα στο έκαση. Το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 5 για τα άλλα όργανα. Θα δώσουμε το λόγο στην ΕΛΓΑ, αλλά θέλω να σας πληροφορήσω ότι το καλοκαίρι μας υποβλήθηκε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο έτοιμα επιτάχυνσης της εξέτασης του διορθωτικού προϋπολογισμού 4. 4. Και μετά από διαβούλευση με τους συντονιστές και συντονίστριες δέχτηκα εξ ονόματος της Επιτροπής μας εφόσον βέβαια θα το δεχτείτε κι εσείς το αίτημα αυτό. Γιατί, διότι εδώ πρόκειται για πρόσθετα μέσα που θα διατεθούν στο Frontex, κονδύλια, που χρειάζεται, πρέπει να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της Αραβικής Ανοίξεως. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ κανονικά ήταν το χρονοδιάγραμμα όπως ήταν θα αλλάξει ως εξή. Στις 13 Σεπτεμβρίου ο διορθωτικός προϋπολογισμός 4 πρέπει να έχει εγκριθεί χωρίς τροποποίηση από το Συμβούλιο. Στις 14 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι λίγη η διορία κατάθεση τροπολογιών από εμά. 22 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και έγκριση στην Ολομέλεια, τη δεύτερη Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Αυτό βέβαια προϋποθέτει πρόσθετη προσπάθεια από εμά ώστε οι τροπολογίες να κατατεθούν μόνο στην αγγλική. Αν και είμαι Γάλλος, είμαι αναγκασμένος να κάνω αυτή την πρόταση, είναι μια θυσία που κάνουμε. Τώρα για τον 5, Έλγα. Ευχαριστώ. Ο διορθωτικός προϋπολογισμός ε, για 5 αφορά τα σχέδια ε, για τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Αυτή η υποπτική υπηρεσία προαπαιτεί ε, μεταμόρφωση ε, θέσεων AD14 σε AD15. Οι πληροφορίες που λάβαμε καταδεικνύουν ότι η αναβάθμιση των θέσεων αυτών είναι όντως δικαιολογημένη. Ωστόσο, ο κανονισμός προβλέπει ότι η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει τέτοιους διορθωτικούς προϋπολογισμούς αν είναι ε, αν υπάρχουν συνθήκες μη προβλέψιμες και μη αποτρέψιμες. Δεν ε, βλέπω ότι υπάρχει κάποιος ε, πιεστικός λόγος να γίνει αυτή η αναβάθμιση. Αυτό μπορεί να γίνει στα πλαίσια του προπολογισμού 2012 και άρα πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να δεχτούμε τις τροποποιήσεις στην παρούσα φάση για να αποφύγουμε να γίνονται αντιορθωτικοί προπολογισμοί για πολύ μικρές αλλαγές. Αυτό για την πρώτη μεταφορά τώρα για το θέμα του EEAS που θα ήθελε να μετατραπούν 40 προσωρινές θέσεις σε μόνιμες. Πρόκειται για μία απόφαση 12-10 του Συμβουλίου που αναφέρει ότι όταν η υπηρεσία EEAS φτάσει στην πλήρη ισχύ του θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι μόνιμες θέσεις. Θέλει λοιπόν ο οργανισμός να υπάρξει αυτή η μετατροπή. Και η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιείται είναι ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να προβλεφθούν οι βαθμοί των νεοπροσληφθέντων όταν ξεκίνησε ο οργανισμός. αυτό θεωρείται ότι είναι ένα κλασικό πρόβλημα στην φάση σύστασης ενός οργανισμού. Και ο, ο ΙΕΣ χρειάζεται και επίσης ένα σχέδιο για α, Όλα αυτά συνεπάγονται 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, δεν χρειάζονται νέα κονδύλια για τις αλλαγές αυτές. Όλα αυτά έχουν ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό το 2012. Και στην τελευταία συνεδρίαση της ομάδας μας, της Επιτροπής μας, ε, είχα εκφράσει σχετικές ε, αμφιβολίες για τις αλλαγές αυτές. Αυτό το έχει συζητήσει και η Επιτροπή ΑΦΕΤ, αλλά το έχουμε συζητήσει και στα πλαίσια του προπολογισμού για το 2012. Υπάρχει σύνδεσμος με την συζήτηση για τον προπολογισμό 2012. Θα ήταν περίεργο αν γινόταν αυτός ο ρυθμικός προϋπολογισμός και η ΑΦΕΤ παράλληλα ε, αποφάσιζε να περιορίσει τον αριθμό των μόνιμων θέσεων για τον EEAS. Αυτά θα εγκριθούν την επόμενη Δευτέρα. Εγώ θα ήθελα τουλάχιστον μια επικριτική προσέγγιση, αν θέλετε, στο σχέδιο αυτό του EEAS για την ε, μετατροπή του πέμπτου προϋπολογισμού. Θέλουμε να ζητήσουμε και πιο πολύ διαφάνεια σε ό,τι αφορά την πολιτική για το προσωπικό των οργανισμών αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ζουζέν Μανουέλ Φερνάντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τι αμφιβολίες που εξέφρασε η συνάδελφο, η Ελκα Τρίπελ, σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά που ανέφερε και παρεπιπτόντω να την συγχαρώ για την δουλειά που έχει κάνει γιατί φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητο να γίνονται τέτοιοι έλεγχοι Υπάρχει μια δυσανάλογη ιεραρχία σε σχέση και με, άλλους, ε, με άλλα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά τις θέσεις, δηλαδή AD 14, 15 και 16. Στον ε, EEAS υπάρχουν υπερβολικά πολλά άτομα στις υψηλές αυτές θέσεις σε σχέση με άλλους οργανισμούς. Είναι πολλές οι θέσεις AD ε, 14 έως 16 σε ποσοστά σε σχέση με, άλλες, ε, με άλλα θεσμικά όργανα. Και είναι σημαντικό να ξέρουμε και να καταλάβουμε αν αυτό πραγματικά είναι δικαιολογημένο. Ιδάλλως, μπορεί να καταλήξουμε να αντιμετωπίζουμε τον EES με διαφορετικό τρόπο και δεν βλέπω γιατί. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομος για τα δύο άλλα θέματα. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στην αρχή, να σας πω την αλήθεια, δεν ε, θεωρήσα ότι υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί αυτό αφορούσε μόνο μία θέση, αλλά καταλαβαίνω και το δέχομαι αυτό που λέει η εισηγήτρια σε ό,τι αφορά την σωστή προσέγγιση. Και θεωρώ ότι ναι, όντω, ίσω να μην υπάρχει ανάγκη επικύρωση στην παρούσα φάση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπηρεσία εξωτερική δράση, το e e Νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο και θα ήθελα να παρακαλέσω την εισηγήτρια να μας δώσει πιο πολλές πληροφορίες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες πρόσληψης που χρησιμοποιούνται. Merci. Ευχαριστώ. Ακούσατε λοιπόν ποια είναι η θέση της εισηγήτριας και των άλλων ομιλητών. Να σας υπενθυμίσω ότι το Συμβούλιο θα αποφανθεί στις 12 Σεπτεμβρίου. Και θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι η απάντησή του στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διορθωτικό προπολογισμό υπαριθμών 5. Σας ευχαριστώ και τώρα συνάδελφοι να πάμε στο σημείο της κυρίας Ματέρα. 14 δηλαδή, το σημείο 14. πριν κοιτάξουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προσαρμογή του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρουσιάσω στους συναδέλφους ε, τέσσερα τέσσερις νέες τροπολογίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την προσαρμογή στην ε, τροπολογία. Η πρώτη τροπολογία από την Πορτογαλία. Θέλουμε να υποστηρίξουμε 600 ε, απολυθέντες από τη Σάντα Μαρία Νταφέρα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ε, τομέα της βιομηχανικής παραγωγής υποδημάτων. Πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος έχει πληχθεί πολύ έντονα από την κρίση μετά στη Δανία στην περιοχή, στην περιφέρεια Μίτλαντ. 325 ε, απολυθέντες από έξι επιχειρήσεις, οι οποίοι απασχολούνταν στον τομέα της μηχανολογίας των αερογεννήτριων. 3,44 δισεκατομμύρια ευρώ ζητούν. Τρίτη, ε, τρίτο αίτημα 778 ε, ε, υπάλληλοι από τη Γερμανία στην Τούσελντορφ στον τομέα της παραγωγής οχημάτων. Να σας υπενθυμίσω ότι το τομείο αυτό δεν υποστηρίζει μόνο απολυθέντες λόγω της παγκοσμιοποίησης, όχι, υποστηρίζει και εργαζόμενους που πλήττονται από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Από την, τον Düsseldorf λοιπόν. Εδώ, το εδώ λοιπόν στον Düsseldorf ε, αφορά 7,34 δισεκατομμύρια ευρώ. Τελευταίο αίτημα από τη Γαλλία. Μία τεράστια βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, μία από τις πιο μεγάλες βοήθειες, ένα από τα πιο μεγάλα ποσά ύψους ε, συγγνώμη, προς υποστήριξη των ε, για εργαζόμενους του Ρενό 3.580 ε, εργαζόμενοι το ποσό που ζητούν αφορά 24,49 εκατομμύρια Η προθεσμία είναι σήμερα στις 3 και η έγκριση στην Ολομέλεια προβλέπεται, αν όλα πάνε καλά φυσικά, προβλέπεται λοιπόν για τη δεύτερη εμ, σύνοδο του Στρασβούργου του Σεπτεμβρίου. Ολοκλήρωσα λοιπόν αυτά που είχα να πω. Να ρωτήσω αν θέλετε να τα ψηφίσουμε. και έχουμε και τέσσερα αιτήματα από τις κάτω χώρες τα οποία θα πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι έτοιμος, αν θέλετε και πρόθυμος να τα ψηφίσουμε αυτά. Τι γίνεται με αυτά που μας παρουσίασε για πρώτη φορά σήμερα η κυρία Ματέρα. Θέλετε το λόγο μήπως. Α, μάλιστα, ορίστε. Euh, Θα ήθελα να δηλώσω στην κυρία εισηγήτρια ότι καταθέσαμε τροπολογίες. για την κινητοποίηση του ταμείου αυτού, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και το αίτημα έχει διατυπωθεί πριν από δύο χρόνια ήδη και πάνω. Εμείς έχουμε έρθει σε επαφή με 887 απασχολούμενους στο εργοστάσιο αυτό και δεν ζήτησαν όλοι να επωφεληθούν από το Ταμείο διότι είχαν δεχτεί να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα αλλά τελικά εδώ και 18 μήνες πριν την συνταξιοδότησή τους βρίσκονται χωρίς κανένα μισθό και είναι ιδιαίτερα δύσκολο για αυτούς να βρουν και κάποια άλλη δουλειά. Τους μειώνεται δε και η σύνταξη που θα τους χορηγηθεί ήδη. Γι' αυτό με τις τροπολογίες μας ζητούμε κάποιες αλλαγές. Και ήθελα να το ξέρει η συγγήτρια. Ευχαριστούμε πολύ. Προτείνω να ψηφίσουμε τις τέσσερις Ολλανδικές προτάσεις που τις έχουμε ήδη συζητήσει και παρά την απουσία ορισμένων Ολλανδών μας συναδέλφων, από τους ενεργότερους μάλιστα στην Επιτροπή μας, Λέω λοιπόν να ψηφίσουμε. Έχω κατάλογο τροπολογιών που τα αφορά και τα τέσσερα θέματα. Ναι, έχετε τον κατάλογο ψηφοφορίας ελπίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, για το α κεφαλαίο, τροπολογία 1, η 3 υπέρ, υπέρ, κατά. Α, μάλιστα. Ξανά υπέρ. Κατά. 10 εγκρίνεται τροπολογία 2 Αλβάρο εισηγήτρια κατά υπέρ κατά μεγάλες ομάδες βλέπω αποχές απορριψετε 3 εισηγητής κατά εισηγήτρια κατά υπέρ της τροπολογίας 3 για την παράγραφο 2 Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τέσσερα. Αλβάρο, η συγκίτρια υπέρ υπέρ. Πολύ. Κατά. Λίγοι. Αποχές. Καμία. Εγκρίνεται. Πέντε. η συγκίτρια κατά υπέρ. Κατά. περισσότεροι. Απορρίπτεται. 6 Αλβάρο εισηγήτρια κατά υπέρ. Κατά. Πολλοί. Αποχές. Ουδήσει. Οι πολλοί κερδίζουν απορρίπτεται. 7 εισηγήτρια κατά υπέρ. Α, ωραία. 1, 5, 7, 10, 14, 13, 15. 16. Κατά. Α. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Τελική ψηφοφορία υπέρ. Υπέρ. Αυτό Κατά. Αυτό. Αποχές. Με μία αποχή λοιπόν. Εγκρίνεται. Συγχαίρουμε την εισηγήτρια και προτείνω τώρα να ψηφίσουμε μαζί και αμέσως όλες τις σχετικές μεταφορές. Δηλαδή 13, 14, 15 και 16. Υπέρ. Συνήθως οι ίδιοι πρέπει να είναι. Κατά. Οι ίδιοι αποχές. Οι ίδιοι. Τα ίδια με πριν λοιπόν εγκρίνεται. Συγχαίρουμε την εισηγήτρια και θα πληροφορήσουμε σχετικώς τους Ολλανδούς μας συναδέλφους για την ψηφοφορία αυτή. Είμαι πεπισμένος ότι θα χαρούν ιδιαίτερα. Και μάλιστα και σε άλλες ψηφοφορίες. Λοιπόν, τώρα επανερχόμαστε στο σημείο 7 και στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξής μας διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα γίνουν και άλλες ψηφοφορίες, αλλά μετά, μετά, μετά, είναι ευθέτω χρόνο. Για το πολιετές πλαίσιο λοιπόν, αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ γρήγορα, δεν προτείνω να το ξανασυζητήσουμε επί της ουσίας. Είναι πληροφόρηση βασικά. Χάρη στη σταθερότητα του Κοινοβουλίου και ιδίως του Προέδρου Μπούζεκ και της Επιτροπής μας, στη διαπραγμάτευση του προπλογισμού του 11 καταφέραμε μεταξύ άλλων οι προεδρίες του Συμβουλίου, οι διαδοχικές προεδρίες, να δεχτούν την εφαρμογή μιας διαδικασίας που επιτρέπει πραγματική ανταλλαγή απόψεων, δηλαδή διαπραγμάτευση μόνιμη για τις δημοσιονομικές προοπτικές καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου για το θέμα αυτό. Αυτό είναι πρωτοφανές σε σύγκριση με την προηγούμενη κατάσταση. Η Πολωνική Προεδρία, μάλιστα, έφτασε μέχρι του σημείου να προσκαλέσει αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας να συμμετάσχει σε άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για να συζητήσει μεταξύ άλλων και τις δημοσιονομικές προοπτικές και έχουμε εκεί στείλει τέσσερις συναδέλφους που πήγανε και συμμετέσχον μαζί με τα μέλη του Συμβουλίου, του υπουργού δηλαδή. Και έκαναν μία γραπτή αναφορά που θα μοιραστεί σήμερα τώρα ή ηλεκτρονικά. Οι ίδιες οι διαπραγματεύσεις λοιπόν θα αρχίσουν επισήμως την επόμενη Δευτέρα επισήμως επίσημη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων και σύμφωνα με αυτή την καινούργια διαδικασία προηγουμένως και μετά θα γίνει συνάντηση αντιπροσωπείας του Συμβουλίου από τρεις υπουργούς των τριών προεδριών με αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου. Άρα πριν το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, πριν να συζητήσει το θέμα αυτό, το Συμβούλιο, αντιπροσωπεία του θα συναντήσει αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου και μετά τις εργασίες του Συμβουλίου, αμέσως μετά, η ίδια αντιπροσωπεία του Συμβουλίου, το τρίο λοιπόν, η Πολωνική Προεδρία, ο Δανός Υπουργός και ο Κύπριος Υπουργός, θα συναντήσουν την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για ενημέρωση. Αυτό σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ορίσει ποια θα είναι αυτή η αντιπροσωπεία του. Η απόφαση είναι αρμοδιότητα της διάσκεψης των Προέδρων. Γιατί, διότι στην πολιτική συμφωνία που συνήφθη πέρυσι με το Συμβούλιο προβλέπεται περιοδικά τα προβλήματα του προϋπολογισμού, ιδιαίτερα δε η διαπραγμάτευση των δημοσιονομικών προοπτικών, να την χάνουν ενημέρωσης, επιτήρησης ε, σε ανώτατο επίπεδο από τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και τον πρόεδρο της Κομισιόν. Τρεις-τέσσερις συναντήσεις έχουν ήδη γίνει σχετικά, λίγο πολύ άτυπα, πριν αρχίσουν επισήμως οι διαπραγματεύσεις. Άρα οι πρόεδροι των ομάδων και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θεωρούν ότι αυτοί πρέπει, οι ο των πρόεδρων δηλαδή, να καθορίσουν τη σύνθεση της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου. Οι πρόεδροι όμως δεν συμφώνησαν για τη σύνθεση αυτής της αντιπροσωπείας και αποφάσισαν μια προσωρινή σύνθεση που θα εφαρμοστεί την επόμενη Δευτέρα αλλά μόνο την επόμενη Δευτέρα και στην επόμενη τους συνεδρίαση, την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο δηλαδή, θα γίνει η τελική, ο τελικός καθορισμός της σύνθεσης της μόνιμης αυτής αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου. Είναι σχετικά επίγον γιατί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συνεδριάζει κάθε μήνα και η επόμενη του συνεδρίαση θα γίνει τον Οκτώβριο. Η διάσκεψη των Προέδρων λοιπόν αποφάσισε. Εσ η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου την επόμενη Δευτέρα να αποτελείται από τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, την πρόεδρο την Ούτα Χάουκ και τον εισηγητή Ράινερ Μπέγκε. Προσωρινά. Αυτό θα γίνει λοιπόν την επόμενη Δευτέρα. Προσθέτω ότι παράλληλα με την ε, διαπραγμάτευση των δημοσιονομικών προοπτικών και προτάσει του Κοινοβουλίου με βάση την έκθεση της Επιτροπής ΣΟΥΡ προεδρεύοντος του Σαλβαδόρ Γκαρίγκα η Πολωνική Προεδρία δέχτηκε να οργανώσει διάσκεψη μια πρώτη διάσκεψη, θα γίνουν και άλλες δημοσιονομική και για θέματα προϋπολογισμού δημόσια και ανοιχτή όχι μόνο σε όλα τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και στο σύνολο των κυβερνήσεων σε υπουργικό επίπεδο και ιδιαίτερα στο σύνολο των εθνικών βουλών και κοινοβουλίων. Έχουν ήδη σταλεί προτάσεις, προσκλήσεις για τις 20 και 21 Οκτωβρίου. Υπάρχει και προσχέδιο ημερήσιας διάταξης για ανταλλαγή απόψεων και για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και το μέλλον του, πώς θα μπορούσε δηλαδή να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα ανάπτυξη της Ένωσης και για τη χρηματοδότηση του στο μέλλον. Αλλά επίσης, θέμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και για το οποίο μίλησε επίσης η Φραντσέσκα Μπαλτζάνη κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται ο συντονισμός του περιεχομένου των εθνικών προϋπολογισμών με τον ενωσιακό για να επιτευχθούν οι στόχοι του 2020 κλπ. Επ' αυτού λοιπόν πρέπει να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει, δεν είναι θέμα όμως μόνο της Επιτροπής μας, αλλά της διάσκεψης των Προέδρων, γιατί 40 εθνικοί βουλευτές θα συμμετέχουν στις συνεννοήσεις αυτές, δύο ανακοινοβούλιο περίπου. Α, πάνω από 40 λοιπόν. 80, 80. Δεν ξέρω, τέλος πάντων θα δούμε. Δύο τουλάχιστον εθνικοί βουλευτές αναχώρα. Δύο αναχώρα. γιατί σε ορισμένες χώρες υπάρχουν δύο βουλές, άνω και κάτω, και για να εκπροσωπηθεί έτσι η κάθε χώρα και από το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία και από το αντιπολιτευόμενο. Επομένως, η διάσκεψη των Προέδρων θα αποφασίσει τον αριθμό και τη σύνθεση της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου. Πρέπει να κάνουμε σχετικά προτάσεις και στην επόμενή μας συνεδρίαση να προτείνουμε και την ημερήσια διάταξη και τη σύνθεση καθώς και τι αποτελέσματα θέλουμε να πετύχουμε και τι συνέχεια θα δοθεί και επιτήρηση και πώς θεωρούμε ότι πρέπει η διάσκεψη αυτή να συνοδεύει τις διαπραγματεύσεις για τις δημοσιονομικές προοπτικές, αν χρειάζονται βελτιώσεις, αλλά χωρίς να καταστήσουμε τα πράγματα πιο δύσκολα και πολύπλοκα και χωρίς η διάσκεψη αυτή τι να υποκαθιστά την ίδια τη διαπραγμάτευση. Είναι κάτι το καινούριο. Εμείς το προτείναμε βέβαια και πρέπει κάτι να φανταστούμε, να εφεύρουμε τώρα. Θα το δούμε με τους συντονιστές και συντονίστριες και θα κάνουμε προτάσεις στην επόμενή μας συνεδρίαση και μετά θα τις υποβάλουμε στη διάσκεψη των Προέδρων. Μήπως θέλει κανείς να συμπληρώσει τίποτε ήδη από τώρα. Μήπως από τους συναδέλφους που ήταν στο ΣΟΠΟΤ θέλει κανείς να σχολιάσει τίποτα. Εντάχει πρόεδρε, διότι όπως ήδη είπατε εμείς ε, υποβάλαμε ένα σημείωμα το οποίο λάβατε και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να εγκριθεί αυτή η υπόμνηση, αυτό το σημείωμα πριν διανεμηθεί και από όσο γνωρίζω υπήρξε θετική ανταπόκριση και η Πολωνική Προεδρία θέλει το Κοινοβούλιο να είναι παρόν με τους Γκαρίγκα, Φέρμς Γένσεν και δέχτηκε την άποψη των συναδέλφων γνωρίζει πολύ καλά ότι υπάρχουν θέματα καθαρά δημοσιονομικά και δεν μπορούμε παρά να δεχτούμε αυτό το πλαίσιο ανάγκης για να συζητηθούν τα θέματα αυτά και το μόνο που δεν μας ανέφερε η Προεδρία είναι τι θα γίνει κατά πόσο ε, θα προβλεφθεί ένα χρονοδιάγραμμα για τις συζητήσεις με το Κοινοβούλιο. Σήμερα θα λάβετε το σημείωμα των συναδέλφων και μου που παρευρεθήκαμε εκεί σε αυτές τις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Άλλοι που ζητούν το λόγο φαίνεται πως όχι. Σας ευχαριστώ. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης. Το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρατών ήδη έχει συζητηθεί η έκθεση Haglund Ο φίλος μας ο Καλ Χάγκλουντ δεν είναι εδώ, αλλά μπορεί να τον αντικαταστήσει η Αν Γένσεν. Ίσως θα ήταν σκόπιμο, μάλλον μου είπαν ότι προετοιμάζεται μία τροπολογία συμβιβασμού. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα μπορούσε να μας το πει η Αν. Ε, αν έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο κείμενο το οποίο έχετε μπροστά σας για να αποτυπωθούν και οι διαπραγματεύσεις με τους οι εισηγητέ και με τον κύριο Μπέγκε προκειμένου το κείμενο πλέον να συνάδει με την στρατηγική που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Η στρατηγική ποια είναι ότι δεν θέλουμε να χρηματοδοτηθεί το ίτρε από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Και πώς θα το πετύχουμε αυτό. Καταρχάς, ίσως να βρεθούν χρήματα κονδύλια από το περιθώριο. Αυτό θα εξαρτηθεί από τον προπολογισμό του 2011 για την Γεωργία. Κατά δεύτερον, αν δεν επαρκέσουν τα κονδύλια αυτά, θεωρούμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το μέσο ευελιξίας για τα κονδύλια που χρειάζονται. Και για να καταστεί σαφές αυτό, τι θα προτείνει ο Κάρλ. Να γίνει περικοπή του προϋπολογισμού του Ήτρε κατά το ποσό το οποίο θα αφαιρεθεί από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Στη συζήτηση θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξή. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες ε, ε, στον ΙΤΕΡ λόγω του σεισμού στην Ιαπωνία. Να μας πει λοιπόν η Επιτροπή κατά πόσον η κατάσταση αυτή σημαίνει ότι θα αλλάξει ο σχεδιασμός του προϋπολογισμού. Twitter μπορεί να συνεπάγεται αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα. Μπορεί να συνεπάγεται ότι θα ακριβίνει η όλη διαδικασία, αλλά ενδεχομένω και να σημαίνει οι περικοπές το 2012 και 2013 αποταμιεύσεις. Να μα το εξηγήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για να είμαστε όμως συγκεκριμένοι, θα γίνουν κάποιες αλλαγές για να αποτυπώνουν αυτά που σας είπα μια μικρή αλλαγή στην τροπολογία 1. Στην παράγραφο 3, στην παράγραφο 1 στην παράγραφο 3 θα γίνει κάποια αλλαγή στα αριθμητικά στοιχεία. Αναφέρεται ότι το πλαφόν θα πρέπει να αυξηθεί κατά 650 εκατομμύρια το 2012 και 119 το 2013 από ό,τι εκπώνοντας όσα σας είπα την στρατηγική των περικοπών προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση και τα χρήματα να προέλθουν από το Ταμείο Ευελιξίας, από το Μέσο Ευελιξία. Κατά, τέταρτον, κατά τρίτον, α, στην τροπολογία 4, το κείμενο που έχετε μπροστά σας, θα μπορούσε να ερμηνευτεί ότι είμαστε υπέρ του διακυβερνητικού χαρακτήρα. Ασφαλώς και δεν είμαστε, άρα και θα αλλάξουμε το κείμενο και να λέει ότι θα χρηματοδοτηθεί από τα κράτη-μέλη και όχι από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, θα αλλάξει και θα γίνει και θα γίνει ε, θα χρηματοδοτηθεί εκτός των πλαφών του MFF. Στην τροπολογία 5 δεν έχω τίποτα καινούργιο να σας αναφέρω. Στην τροπολογία 6 ε, έχουν γίνει αλλαγές στα αριθμητικά στοιχεία και πάλι έχουμε αριθμιστικά στοιχεία τα οποία αναφέρουν ότι το ανώτατο ποσό από το πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να είναι 270.000 Διαγράφουμε λοιπόν τα 46 εκατομμύρια. Και επίσης παρακάτω φεύγουν και η ενέργεια και η έρευνα. δηλαδή από 1.748 εκατομμύρια, το ποσό πλέον είναι 2 εκατομμύρια, 2 δισεκατομμύρια 108 εκατομμύρια. Αυτές είναι οι αλλαγές για τις περικοπές. Όλα αυτά γίνονται για να εξασφαλιστεί ότι τα χρήματα, τα κονδύλια δεν θα προέλθουν από το έντομο πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά θα προκύψουν από όσα δεν θα απανηθούν στο πρόγραμμα για τη γεωργία για το 2011 ή από το μέσο ευελιξίας. Αυτά είναι λοιπόν τα δύο στοιχεία. Όχι από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και κατά δεύτερον να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον έχει γίνει, έχουν γίνει αλλαγές σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό για τον ίτερ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Άρα θα γίνει κοινή συζήτηση με το σημείο 11 που αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσαρμογή του πλαισίου, του πολιετούς χρηματοοικονομικού πλαισίου. Ο κύριος ε, Μπέγκε είναι εισηγητής. Η Χάγκλουντ και Μπέγκε συνεργάστηκαν διότι το ίτερ αποτελεί, αποτελεί μάλλον το ίτερ αφορά και τον προπολογισμό 2012 ε, και αφορά την έκθεση Haglund. Ράιμερ, θέλεις κάτι να προσθέσεις. Yeah, uh, ο κύριος ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν είναι εδώ η συγητής. Θα τον ευχαριστήσω όμως για την έκθεση και για την ε, εμπέσμευσή του και για τις συζητήσεις που έκανε με τους κοιόδης. Και φυσικά συμφωνούμε ότι θα πρέπει σκοπός μας είναι να προστατέψουμε το πρόγραμμα πλαίσιο 7, το 7 πρόγραμμα πλαίσιο. Θα χρησιμοποιηθεί και θα δαπανηθεί πλήρως φέτος, άρα ίσως να μην υπάρχει τίποτε επιπλέον. Πού θα βρούμε όμως τα κονδύλια να χρησιμοποιήσουμε τον φάκελο για τον Ίτερ. Αυτά που είπε η συγκήτρια, ο εισηγητής. Εγώ νόμιζα ότι είχαμε συμφωνήσει για τα αριθμητικά στοιχεία, για τα ποσά σε ό,τι αφορά για τον Ίτερ. Απλά δεν είχαμε συμφωνήσει για το πώς θα βρούμε τα κονδύλια αυτά. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να φέρουν το κόστος αυτό. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, όπως προτείνει ο εισηγητής, το μέσο ευελιξία. Υπάρχουν άλλες λύσεις. Να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, τα περιθώρια. Υπάρχουν και άλλες λύσεις, αλλά θα πρέπει να πούμε στην παρούσα φάση ότι δεν θέλουμε μεν να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα πλαίσιο, αλλά να δώσουμε και τις άλλες λύσεις και οι σοσιαλδημοκράτες θα υποβάλουν κάποιες προτάσεις σε ό,τι αφορά τη διατύπωση. Ευχαριστώ. Έχουν ζητήσει πολύ το λόγο. Σαβάλ. Απλώς θα ήθελα να σας ε, ε, δώσω μία πληροφορία. Μιλήσαμε για περικοπές του εβδόμου ου προγράμματος πλαισίου πολλές φορές για να χρηματοδοτήσουμε το ίτερ. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι η πορεία εκτέλεσης του εβδόμου ου προγράμματος πλαισίου. Δηλαδή υπάρχουν τα, τα χρήματα αυτά για την ε, χρηματοδότηση του ΙΤΕΡ και η Επιτροπή μας λέει ότι όχι μόνο δεν θα υπάρξουν χρήματα, αλλά επειδή έχουν γίνει περίκοπες, ίσως χρειαστεί και μία μεταφορά πιστώσεων. Και λέει ότι η κατάσταση των πληρωμών το 2011 είναι πιο δύσκολη εξαιτίας των περικοπών και αυτό ίσως θα χρειαστεί συνολική μεταφορά του προϋπολισμού 2011 προς το τέλος του έτους για την χρηματοδότηση. Σε σχέση με την πρόταση προϋπολογισμού για το 2012, το ποσό αφορά τον αρχικό προγραμματισμό και θα εκτελεστεί κατά 100%. Άρα υπάρχει πρόβλημα εκτέλεσης διότι δεν υπάρχουν χρήματα, αρκετά χρήματα στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Γι' αυτό ακριβώς δεν θα έπρεπε να γίνουν περαιτέρω περικοπές στο 7ο πρόγραμμα για να, χρηματο, για να χρηματοδοτηθεί το ίτερ. Η Helga Τρούπελ έχει το λόγο. Ναι, συμφωνώ με τη θέση ότι ο ΙΤΕΡ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το 7ο πρόγραμμα για την έρευνα, αλλά αυτό που θεωρώ ότι είναι πολύ περίεργο είναι να προέλθουν τα κονδύλια από το μέσο ευελιξία. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο κατεπίγουσε ανάγκε σε ό,τι αφορά το μέσο ευελιξία. Και εμεί οι πράσινοι δεν είμαστε γενικότερα υπέρ του ΙΤΕΡ, το ξέρετε, το επαναλαμβάνω. Effectivement, euh, quel que soit le sentiment qu'on peut avoir sur le projet, Πράγματι, το ξέρουμε γιατί η χρήση ενός μέσου ευελιξίας για τη χρηματοδότηση ενός ε, ε, τέτοιου προγράμματος σημαίνει ε, ότι υπάρχει μία λογιστική εφευρετικότητα. Συμφωνώ σε ό,τι αφορά τη μη χρήση του εβδόμου προγράμματος ε, πλαισίου. Ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι υπέρμαχοι του project θεωρούν ότι το 2050 δεν θα έχει προκύψει, δεν θα χρησιμοποιεί, μέχρι το 2050 δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ενέργεια, αυτή την τεχνολογία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους και θα πρέπει να πω στην αν το εξή. Στην Καταράς είδαμε ότι τα κράτη-μέλη κάθε ευρώ που δεν δαπανάτε που εξοικονομείται ε, τα κράτη-μέλη έχουν καταφέρει να περάσει, να επιστρέφεται στα κράτη-μέλη. Άρα, εγώ θα ήθελα τα αποθέματα τα οποία σχηματίζονται, ακόμα και αν είναι μικρά, να μένουν στο project. Θεωρώ ότι αποτελεί ένα συμβολικό, αν θέλετε, μια συμβολική συμβολή για την πραγματοποίηση του project. Ευχαριστώ, κυρία Να πω ότι καταλαβαίνω αυτά που λέτε για το 7ο πρόγραμμα και στο τέλος κάθε προγραμματικής περίοδου φυσικά ανακύπτουν διαρκώς νέες ανάγκες και υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για κονδύλια αφετέρου να προσέξουμε. Να μην ε, αντιμετωπίζουμε το ίτερ ε, ως ένα πρόγραμμα εξαιρετικό αν θέλετε και όχι ως ένα κοινό πρόγραμμα έρευνας. Θεωρώ ότι είναι ένα κοινό πρόγραμμα έρευνας, μακροπρόθεσμο. Και θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προκύψει μία διακυβερνητική ρύθμιση σε σχέση με τον ΙΤΕΡ. Ή για παράδειγμα να επιστραφούν τα κονδύλια τα οποία δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί για την γεωργία στα κρατημέλη και τα κρατημέλη να τα επανεισάγουν χωρίς να έχουμε εμείς ως κοινοβούλιο αν οποιαδήποτε συμμετοχή. Θα πρέπει να είναι ισχυρή τοποθέτησή μα στις διαπραγματεύσει και θα πρέπει φυσικά και εμείς αλλά και οι κυβερνήσει να επαναχωρήσουμε σε σχέση με την αρχική μας θέση προκειμένου να είναι ισχυρή η θέση του Ίτερ. Πολλά ε, ερωτήματα θέσαμε στο Κανταράς και πολλά από αυτά έχουν ε, απαντηθεί εντελεχώς. Άρα όλα όσα κατηγορούσαμε στο παρελθόν περί αδιαφάνειας πρέπει να πούμε ότι βελτιώνονται σαφώς. Και θεωρούμε ότι και στην διεύθυνση, στην διαχείριση υπάρχει μια συνέπεια, μια διαφάνεια και ελπίζω αυτή η τάση να συνεχιστεί. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν την ε, εκπρόσωπο του εισηγητή. Ο Γενικός Γραμματέας είναι αφηρημένος. Έχει πολλές όμορφες γυναίκες γύρω του, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της τραγωδίας της Φουκουσίμα σε σχέση με την προμήθεια εξοπλισμού από την Ιαπωνία για το κέντρο του Κανταράς. Δηλαδή κατά πόσο αυτό θα έχει επιπτώσεις ως προς τις προθεσμίες. Σας υπενθυμίζω ότι ως προς το χρονοδιάγραμμά μας, σε σχέση με την έκθεση αυτή, η προθεσμία υποβολής τροπολογιών στις 12 ε, Σεπτεμβρίου, ψηφοφορία στις 22 στην Επιτροπή, γνωμοδότηση από την Ήτρε που θα ψηφίσει στις 6 Οκτωβρίου και θα περάσει στην Ολομέλεια είτε τον Οκτώβριο 2 είτε τον Νοέμβριο. Δεν είναι ακόμα σαφές. Σας προτείνω να περάσουμε τώρα στο 12 την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε ε, στην ΑΦΕΤ. Ο Γκέραν έχει το λόγο. Ε, yes, this is... Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, είναι μια γνωμοδότηση στην έκταση της Επιτροπής Εκτορικών Υποθέσεων για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία να υπενθυμίσουμε ότι δεν μιλάμε μόνο για την κατάσταση που αφορά τη Μεσόγειο, την Αραβική Άνοιξη. Όχι, μιλάμε αναθεώρηση, για αναθεώρηση του μέσου για την πολιτική γειτονία και προς ε, ε, τον Νότο και προς τον Ανατολάς. Ανταποκρινόμαστε λοιπόν στην έκθεση της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Φυσικά εστιαζόμαστε σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικά ζητήματα. Δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνουμε πολιτικά επιχειρήματα που έθεσε η Επιτροπή ΑΦΕΤ, αλλά θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν μπορούμε να εστιαζόμαστε μόνο στο νότο, παρόλο που είναι πιο έντονη η κατάσταση εκεί. Καταρχάς, λοιπόν, θέλουμε να τονίσουμε το εξή, Κοιτάμε στα πλαίσια του προϋπολογισμού του 2011 και ένα διορθωτικό, μια διορθωτική επιστολή για τον προϋπολογισμό 2012 κοιτάμε την μεταρρύθμιση αυτού του μέσου ή μάλλον τη δημιουργία ενός καινούριου μέσου και ένα από τα βασικά στοιχεία είναι ότι θα πρέπει να βρούμε μια στρατηγική η μαλλον τη δημιουργια ενος καινουργιου μεσου και ενα απο τα βασικα στοιχεια ειναι οτι θα ισχύει για όλους τους τομείς που μας απασχολούν. Δυστυχώς το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων πριν από το καλοκαίρι δήλωσε ότι το θέμα αυτό θα τους απασχολήσει έντονα αλλά θέλουν να αποφύγουν τις επόμενες ε, μακροπρόθεσμες προπτικές από πλευράς ε, της Επιτροπής μας θα πρέπει να αποφύγουμε τις αλεπικαλύψεις γιατί έχουμε φυσικά την Ένωση για την ε, Μεσόγειο για παράδειγμα θα πρέπει να βρούμε τον σωστό τρόπο για να μην υπάρχουν ε, αλληλεπικαλύψεις. Ένα από τα βασικά ζητήματα που θα μας απασχολήσουν και πρέπει να μας απασχολήσουν είναι το ποια μέσα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αφενός υπάρχει ο προπολογισμό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει όμως και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Θα πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος του κάθε οργάνου και επίσης να συγκρίνουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το ρόλο των κρατών μελών. Αυτό αποτέλεσε σημαντικό πολιτικό πρόβλημα στο παρελθόν και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Πολλά κράτη-μέλη έχουν συμφέροντα, ιδιαίτερα στην ε, νότια διάσταση της πολιτικής γειτονίας. Η Γαλλία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τα συμφέροντά τους, τα ξέρουμε όλα αυτά. Θα πρέπει να είναι συντονισμένη η ευρωπαϊκή πολιτική και από πολιτικής άποψης, αλλά και για πολιτικούς λόγους για να αποφύγουμε αλληλεπικαλύψεις, να μην έχουμε αντιφατικά μέσα. Επίσης υπογραμμίζουμε ότι ναι μεν υπάρχει η πολιτική γειτονία, αλλά σε αυτήν εντάσσεται και η χρηματοδότηση της Παλαιστινιακής Αρχής, που όπως ξέρετε είναι πολύ αμφιλεγόμενη εδώ και πολλά έτη. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε και μια μακροπρόθεσμα στρατηγική και για αυτό το τομέα. Η Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα ε, αντιμετώπιζαν τη χρηματοδότηση της Παλαιστινιακής Αρχής ως κάτι το βραχυπρόθεσμο για να ασκούν πίεση στους εταίρους, για να ζητούν πολιτική πρόοδο από τους πολιτικούς μας εταίρους, με, αν θέλετε εκβιάζοντας κάπως. Θεωρώ ειλικρινά ότι αυτό δεν έχει λειτουργήσει ως στρατηγική Χρειαζόμαστε μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση της ΑΝΔΑ και της Παλαιστινιακής Αρχής. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο εντάσσεται απαραίτητα αυτό στην έκθεσή μας αυτή, αλλά θα ήθελα να θέσω την ερώτηση αυτή προς την Γενική Διεύθυνση για τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έγινε μια συζήτηση για τη χρηματοδότηση της Παλαιστινιακής Αρχής, για τη Μεσόγειο και μας είπε ο κύριος Ζαν ότι είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις της Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 2012 που έχουν γίνει περικοπές κατά ένα τρίτο. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Ζαν κατά πόσον έχει κάποια συγκεκριμένη ιδέα για το τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση του Άνδρα και της Παλαιστινιακής Αρχής σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2012 ανέφερα και τα προβλήματα που έχουμε με την ανατολική και νότια διάσταση της πολιτικής γειτονίας, γιατί φυσικά τώρα όλη η επικέντρωση είναι στο νότο. Κατά το παρελθόν πάντα τονίζαμε ότι το 1 τρίτο θα πήγαινε στην ανατολική γειτονία και το 2 τρίτα στην νότια γειτονία. Θα πρέπει φυσικά να υπάρχει μια η ισορροπία. Η ισορροπία αυτή φυσικά θα πρέπει να εξελίσσεται ε, με την πάροδο του χρόνου και λόγω των ε, εκάστοτε αναγκών και λόγω της εκάστοτε πρόοδου. Θα πρέπει να βρούμε όμως μια σωστή ισορροπία, να μην ξεχνάμε παρά τον πιεστικό χαρακτήρα των εξελίξεων ε, στον Νότο. Μην ξεχνάμε ότι οι χώρες προς Ανατολάς είναι χώρες που προσδοκούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μελλοντικά Και κάτι άλλο που ξεχνάμε είναι η δυνατότητα των όμορων χωρών να συμμετάσχουν σε κάποια προγράμματα, εξωτερικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια από αυτά τα προγράμματα, από αυτούς τους οργανισμούς είναι ανοιχτά για συμμετοχή από τρίτους εταίρους και υπάρχει και ένας κίνδυνος, ιδιαίτερα με την πολιτική προσοχή που έχει στραφεί στην περιοχή της Μεσογείου. Πολλές ιδέες ανακύπτουν, πολλές ιδέες για χρηματοδότηση. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε έναν περιορισμένο αριθμό προτεραιότητων, όχι μόνο μεγάλα project, γιατί φυσικά πολιτικός πόσο είναι σαφές ότι είναι πολύ σημαντικό να χρηματοδοτηθεί η κοινωνία των πολιτών, οι περιφερειακές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι. Άρα είμαστε υπέρ των περιορισμένων, του περιορισμένου αριθμού project, αλλά να μην είναι απαραίτητα μεγάλα αυτά τα project. Κάτι άλλο πολύ αμφιλεγόμενο και θα ήθελα να ακούσω και εδώ τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κατά πόσο έχει σημειωθεί πρόοδος. Ξέρετε ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής πρότεινε πακέτο 1,24 δισεκατομμυρίων για την πολιτική γειτονία για το τρέχον και τα δύο επόμενα έτη. Ένα μεγάλο μέρος θα χρηματοδοτηθεί από, τις, ε, από την Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων το 1 πέμπτο. Αλλά ως τώρα, από τις απανές αλλά ως τώρα δεν έχει βρεθεί μια συγκεκριμένη λύση, δεν έχει προταθεί κάτι συγκεκριμένο. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, ή θα χάσουμε το 1 πέμπτο του προγράμματος. Τι προτείνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούν να μας πληροφορήσουν για τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπάρχουν εναλλακτικέ. Και τι θα γίνει άμα δεν υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση. Πού θα το βρούμε αυτό το 20% το 1 πέμπτο. Το πρώτο σχέδιο θα το παρουσιάσουμε κατά βάση σε δύο εβδομάδες. Μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου έχουμε προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών και ψηφοφορία στην Επιτροπή μετά. Έχουμε λοιπόν ένα μήνα ακόμα εδώ στην Επιτροπή για να υποβάλουμε τροπολογίες για να συζητήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα Γκόραν, ήταν πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και με τη συγκυρία που σημειώνεται εδώ στο νότο της Μεσογείου έχει γίνει ακόμα σημαντικότερο. Λοιπόν, ο ζητητής κατέθεσε, έθεσε ορισμένα ερωτήματα στην Κομισιόν και εκείνη ακριβώς τη στιγμή που τα έθετε αναγκάστηκε να φύγει ο Γενικός Διευθυντής αλλά υπάρχει ο Διευθυντής. Μπορείτε να απαντήσετε ήδη από σήμερα στα δύο κύρια ερωτήματά του το ένα για τις πιθανές νέες προτάσεις σας για τον προϋπολογισμό του 12 και το άλλο για τις πιθανές νέες χρήσεις της ΕΤΕ, κύριε Διευθυντά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ορίστε ορισμένα στοιχεία. Για την Παλαιστίνη, το η διορθωτική επιστολή υπαριθμών 1 μιλάει και γι' αυτό και από ό,τι συζητήσατε και εσείς φαίνεται ότι δεν γίνεται κατανομή αναχώρα αλλά μια διαφοροποιημένη κατανομή βάσει των προόδων που έχουν σημειωθεί με βάση προκαθορισμένα κριτήρια. Η Παλαιστίνη λοιπόν είναι τμήμα της γενικότερης αυτής περιφέρειας και σίγουρα είναι από τα θέματα που θα συζητηθούν στη δημοσιονομική διαδικασία, στη διαδικασία εξέταση του προπολογισμού του 12. Δεν υπάρχουν καινούργιες επίσημες προτάσεις της Κομισιόν για τον προϋπολογισμό που να αφορούν συγκεκριμένα το θέμα. Ούτε πρόκειται να γίνουν. Όσο για τα λεγόμενα reflows από την προς την ΕΤΕ αντιμετωπίζουμε ακόμη κάποιο πάγωμα της κατάστασης από το Συμβούλιο και η Κομισιόν θεωρεί ότι η προηγούμενη της πρόταση παραμένει σωστή γιατί υπάρχουν χρήματα για τα οποία δεν χρειάζεται να πληρώσουν τα κράτη. Θα μπορούσαν να προσθεθούν βέβαια νέα ταμεία, αλλά αυτό δεν χρειάζεται νομίζω νέα κονδύλια, γιατί δεν είναι, θα ήταν ό,τι το αποτελεσματικότερο. Η θέση μας λοιπόν είναι να διατηρήσουμε, να συνεχίσουμε την πίεση για να προσπαθήσουμε να συμφιλιώσουμε, να συνδυάσουμε τις πολιτικές δηλώσεις που γίνονται με τις υποσχέσεις που είχαν γίνει προς τα κράτη της περιφέρειας αυτής χρησιμοποιώντας μάλιστα ε, ένα εργαλείο που δεν χρειάζεται να ε, πληρωθεί από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστούμε. Παρακολουθούμε όλοι τι γίνεται στην Παλαιστίνη και ιδιαίτερα τι θα γίνει σε δύο εβδομάδες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ όπως ξέρετε, η Παλαιστινιακή Αρχή αποφάσισε να ζητήσει εκεί επίσημα την αναγνώρισή της από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως ανεξαρτήτου κράτους. Πράγμα που οδήγησε την Ένωση να προσπαθήσει να δημιουργήσει μια κοινή θέση επ' αυτού. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Και απαιτεί, θα απαιτούσε κάτι τέτοιο θα πετούσε λέγω μία κοινή απάντηση από τα κράτη που ανήκουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας ή όπως λέγανε παλιά τις δυτικές δυνάμεις τις μεγάλες δυνάμεις μάλλον βέβαια αν βρεθεί κάποιος τέτοιος συμβιβασμός μπορεί κανείς να φοβηθεί μήπως χώρες σαν τις Ηνωμένε Πολιτείε μειώσουν τη χρηματοδοτική τους συμβολή, τη βοήθεια. Αν αντίθετα υπάρξει πλήρης αποτυχία της πρωτοβουλίας αυτής, τότε υπάρχει φόβος να χρειαστεί χρηματική αντιστάθμιση, αποζημίωση. Πάντως υπάρχει αυτή η ημερομηνία και όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας θα χρειαστεί να πληρώσουμε παραπάνω. Να το προσέξουμε λοιπόν ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε, δεν ζήτησε κανείς το λόγο. Ευχαριστούμε τον εισηγητή που υπενθύμησε και το χρονοδιάγραμμα. Κανονικά η γνωμοδότησή του θα είναι έτοιμη για τις 22 Σεπτεμβρίου, 12 Οκτωβρίου λίγη διορία κατά τροπολογιών και 7 Νοεμβρίου θα εγκρίνουμε εμείς. Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Τώρα θα έλεγα να περάσουμε στο σημείο 13 της κυρίας Βέρτμαν για το σχέδιο τροποποίησης μιας οδηγίας restructuring the community framework κλπ. Κυρία εισηγήτρια, Παρακαλώ να είστε λίγο σύντομοι γιατί έχουμε και ψηφοφορίες. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, ναι. Αγαπητοί συνάδελφοι και πριν το καλοκαίρι σας ε, παρουσίασα πώς είχε η κατάσταση για την οδηγία και νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να επικεντρωθούμε στα πλέον σημαντικά. Τι προτείνει βασικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον η φορολογία ενεργειακών προϊόντων να διαρρεθεί σε δύο κατηγορίες καταρχάς βάσει της περιεκτικότητας σε διοξείδιο του άνθρακα και κατά δεύτερον βάσει της ενεργειακής περιεκτικότητας. Και στις ε, συζητήσεις με τους κοιόδης αποφασίσαμε να εξετάσουμε το θέμα αυτό από πλευράς ε, προϋπολογισμού. Το βασικό είναι το εξής, ότι η φορολογία βάσει διοξιδίου του άνθρακα μπορεί να ε, και μπορεί και θα πρέπει να περιλαμβάνει συμμετοχή των ίδιων πόρων. Και εκτός αυτού υπάρχει και η κοινωνική πτυχή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την φορολόγηση των ενεργειακών παρόχων. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανταποκριθεί σε αυτά που έχουμε ζητήσει. Η γνωμοδότηση την έχετε στη διάχυσή σας πλέον ε, και σε όλες τις γλώσσες. Σας παρακαλώ να καταθέσετε την τροπολογίες και να σας ε, ζητήσω το εξής. Αναφέρεται η 22 Σεπτεμβρίου ως ε, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, ενώ είχαμε αναφέρει στην αρχή στις 28 Σεπτεμβρίου. Τι ισχύει λοιπόν. Και φυσικά καλωσορίζω και σχόλιά σας προκειμένου να είναι αρκετά ανιαία η γνωμοδότηση και να την στηρίξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ήσασταν σύντομοι και ακριβείς. Ως προς τις προθεσμίες, έχουμε προβλέψει τις 22 αν υπάρξει πρόβλημα θα σας το πω. Η κυρία Καρβάλιο ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κυρία Βέρτμαν για την εργασία της, αλλά στο ΕΛΚ ανησυχούμε ως προσωρισμένες τροπολογίες γιατί θεωρούμε ότι δεν σχετίζονται ε, με θέματα της δικής μας Επιτροπής, αλλά της ΕΚΟΝ ή της ΙΤΡΕ. Ένα δεύτερο θέμα όπως είπε και η συγγήτρια, είναι το εξής. συνδέουμε το θέμα των ιδίων πόρων με το θέμα της ε, φορολόγησης του διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό έχει συζητηθεί κάπως διαφορετικά. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ε, σίγουροι ότι δεν δημιουργούμε εντροπία στο σύστημα. Αυτά είναι τα δύο μελήματα του ΕΛΚ επί του θέματος. Ευχαριστούμε. Ελάτε σε επαφή με την κυρία Βέρτμαν για να δείτε κατά πόσο μπορείτε να φτάσετε σε μία συμφωνία. Είναι δύσκολο σε αυτό το θέμα να δούμε ποιο είναι το input της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Γιατί πρόκειται ένα θέμα που αφορά και τις εθνικές νομοθεσίες, την εθνική νομοθεσία. Τα προϊόντα ενέργειας και ηλεκτρισμού δηλαδή. Αλλά όπως μας υποενθύμησε και η εισηγήτρια, στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και στην ΣΥΡ είχαμε πει ότι μας ενδιαφέρει η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού με βάση τη φορολόγηση της ενέργειας που μολύνει. Δεν ζητά κανείς άλλο το λόγο. Σας ευχαριστώ. Μου είπα στο μεταξύ ότι η προθεσμία μπορεί να είναι 28 Σεπτεμβρίου, αν το θέλετε. Είναι το ίδιο για σας. Μπορούμε να αφήσουμε την 20η Δευτέρα ως ε, ημερομηνία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, από εσάς εξαρτάται, ό,τι θέλετε. Απλά ήθελα να σας το τονίσω. Ωραία. Κρατάμε την ε, προτινόμενη ημερομηνία και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην τελευταία ψηφοφορία Σας προτείνω να δούμε το σημείο 21, δηλαδή την έκθεση Τζοβάνι Λαβία ως προς τα ειδικά μέτρα για τη γεωργία στις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες της Ένωσης. Πάρτε την κάρτα σας και τον κατάλογο 34. Πάξας ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Η πλειοψηφία απορρίπτεται. 35. Πάξα. Ο εισηγητή είναι κατά. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. 36. Ο εισηγητή είναι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Κύριε ό,τι θέλετε. Υπέρ. Ε, κατά. Κατά με συγχωρείτε. Αποχές εγκρίνεται. Προτείνω να ψηφίσουμε unblock της 36 μέχρι 40. Χάρτονγκ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 41. Πάξας, εισηγητής κατά, υπέρ παρακαλώ. Κατά απορρίπτεται. Το ίδιο τώρα θα κάνουμε από 42 μέχρι και όλη την επόμενη σελίδα και όλη την επόμενη σελίδα μέχρι την 57. Ο κύριος Σαρτόγκ αποσιάζει. Ψηφίζουμε αμπλοκ υπέρ. Κατά. Μεγάλη πλειοψηφία αποχές απορρίπτονται τροπολογίες του εισηγητή. Σας προτείνω να δούμε αν μπλοκ, να ψηφίσουμε την 1, 2, 3 και 4 υπέρ αυτών κατά 5, 7, 7, 7. Εγκρίνονται παρόλα αυτά. 58 Εστέλ Γκρελιέ αλλά υπάρχει και μια προφορική του εισηγητή ο οποίος ζητά εάν ψηφιστεί να θεωρηθεί αιτιολογική σκέψη 36 υπέρ κατά αποχές, μία αποχή εγκρίνεται. 59. Πρόκειται για το ίδιο, προφορική. Έτσι ώστε αυτό το κείμενο να αλλού, υπέρ. Κατά. Αποχές, ίδια πλειοψηφία, άρα εγκρίνονται. Έχουμε μία σειρά Χάρτονγκ 5 μέχρι το τέλος της σελίδας, μέχρι το, μέχρι το 34, τροπολογία 27, on block, υπέρ, ο εισηγητής είναι κατά. Κατά, σχεδόν όλοι, αποχές απορρίπτονται. Τώρα φτάνουμε στην τροπολογία συμβιβασμού για τη σύμπτυξη των τροπολογιών 28 και 31 του κυρίου Πάξας και της κυρίας Γκρελιέ. Άρα συμφωνούν φαντάζομαι η Πάξας και Γκρελιέ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Πέντε. Αποχές Άρα εγκρίνεται. Άρα ψηφίσουμε την 29 Αρτόγκ υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 Γκρελιέ. Ο εισηγητής είναι κατά. Υπέρ. Α, οι σοσιαλιστές υποστηρίζουν τον κύριο Γκρελιέ. Κατά. Όσοι δεν είναι σοσιαλιστές λοιπόν. Άρα μειοψηφούν οι σοσιαλιστές. 31 καλύπτεται, 32 ψηφίζουμε υπέρ, ο εισηγητής είναι κατά. Κατά, αποχές απορρίπτεται. 33 γκρελιέ, ο εισηγητής είναι υπέρ, υπέρ παρακαλώ. Κατά, 4 εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης υπέρ κατά 5 αποχές Εντάξει, θα σας υπολογίσουμε. Ωραία, σας ευχαριστώ. Εγκρίθηκε η έκθεση Λαβία τον οποίο και συγχαίρω. 22. Εδώ γίνονται ορισμένες μεταφορές. Voilà, c'est 31. Alors, Sidonia n'est Η Sidonia δεν είναι παρούσα. Αλλά μπορώ να σας πω το εξής. κατά τη διάρκεια του θέρους μας ζητήθηκε γνωμοδότηση κατεπηγόντος για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση λοιμού στη Σομαλία και ιδιαίτερα στο κέρας της Αφρικής. Μιλάμε για 100 εκατομμύρια στις υποχρεώσεις και 50 εκατομμύρια στις πληρωμές. Από το απόθεμα επίγουσας βοήθειας και όταν μας, το, μαζητήθηκε ζητήθηκε κάτι τέτοιο τον Αύγουστο, είπαμε ότι η Επιτροπή Προϋπολογισμών μετά από συμφωνία των συντονιστών θα δεχόταν η Επιτροπή μας αυτή τη διαδικασία υπό την προϋπόθεση της δικής σας σημερινής συμφωνίας. Ποιοι είναι λοιπόν υπέρ αυτής της ε, μεταφοράς. Σας ευχαριστώ. Κατά. Ευχαριστώ. Αποχές. Εντάξει. Ομόφωνα. Γίνεται αποδεκτή αυτή η μεταφορά. Από την άλλη πλευρά ψηφίσαμε τις άλλες μεταφορές για τον προϋπολογισμό φέτος που σχετίζονται, ο Γιάνν Μούλτερ δεν, δεν ήταν εδώ όταν ψηφίσαμε, την βοήθεια λοιπόν σε σχέση σχέση με, τη, με την Ολλανδία ως προς το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Με μεγάλη χαρά λοιπόν εγκρίναμε. Η Χέλγα θέλει κάτι να μας πει. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σύμφωνα με το άρθρο 22 και 24 μιλάμε για τον προπολογισμό του Ευρωπαίου Εποπτή Προστασίας Δεδομένων. Προσπαθούμε ε, σκοπός είναι να μειωθούν ε, ε, τα 50.000 κατά 50.000 ευρώ σε ό,τι αφορά τους παιδικούς και προχρονικούς σταθμούς. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει κάποιο πρόβλημα και γι' αυτό λοιπόν σας στείλω να υποστηρίξουμε αυτή την πρόταση. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Οκ. Okay. Υπέρ της πρότασης της εισηγήτριας, ευχαριστώ. Κατά ένας, αποχές, εγκρίνεται λοιπόν. Ως προς το building policy δεν βλέπω τίποτα. Έκθεση Αλφόνση, έπρεπε να σας το πω εξ αρχής, έχει αναπαιμφθεί, διότι ο κύριος Αλφόνση δεν μπορούσε να είναι παρόν, αλλά τελειώσαμε με την ημερήσια διάταξη. Λύεται η συνεδρίαση αλλά θα ήθελα οι συντονιστές να παραμείνουν και οι συγητές με τις αντίστοιχες γλώσσες. Για τους διερμηνείς θα πούμε σε πέντε λεπτά ποιες γλώσσες θα χρειαστούμε και οι άλλοι θα είναι ελεύθεροι.